Συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Δηλαδή, καλησπέρα αντί για καλημέρα. Να καλωσορίσουμε τον Αντιπρόεδρο Κωνστανσίου. αλλά πριν περάσουμε ε, στον διάλογο με την ΕΚΤ, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να σας ζητήσω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Και μια σύντομη ενημέρωση για τις θεσμικές διαπραγματεύσεις. Ο τριμερής διάλογος της 28 Μαρτίου για τον, ε, για τον κανονισμό του ελέγχου ρευστότητα ήταν ο δεύτερος γύρος με τη συμμετοχή των Επιτροπών Νέα Κολύμπη όπως και συνειδητάμε το πεδίο του κανονισμού, την ανάλυση του κινδύνου και το κατά πόσον ε, θα δεχτούμε τροπολογίες για να διευκρινίσουμε την κάλυψη της αξιολόγησης κινδύνου και την οδηγία κατά του ξεπλήματος βρωμικού Την προσωρινή κράτηση μετρητού ρευστότητας, αυτό θα συζητηθεί στον επόμενο τριμερή διάλογο, αλλά μπορεί να προβλεφθούν εξαιρέσει στο γενικό κανόνα για κάποιες περιπτώσεις που αιτιολογούνται. Επίσης, η ανάγκη να έχουμε ένδικα μέσα που να λειτουργούν και την καλή επικοινωνία μεταξύ αρμόδιων αρχών συμπεριλαμβανομένων των τροπολογιών του Κοινοβουλίου για τη διασύνδεση των ε, δικτύων ε, ενημέρωσης, των βάσεων δεδομένων. Ακόμη υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, ιδίως την περίοδο ε, αποστολής πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, αλλά επιδείχθηκε διαλλακτικότητα και από τις δύο πλευρές και η περαιτέρω αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι απαραίτητη για την ε, αλληλοδιασύνδεση αυτή. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρξει αρκετό χρόνο για την ε, εφαρμογή αυτή τη διασύνδεση και για την τήρηση των δεδομένων και το αν είναι μακρά η διάρκεια ή όχι. Το Συμβούλιο επιμένει στην στάση του. Εμείς θα ελέγξουμε σε επίπεδο κρατών μελών κατά πόσον μπορούν να δείξουν διαλλακτικότητα για τις ποινές. Το Συμβούλιο συμφωνεί με το στόχο να υπάρχει ένα συντονισμένο σύνολο ποινών και κυρώσεων για να μην υπάρχει άγρα δικαιοδοσία και να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση. Η επόμενη και ελπίζουμε τελική φάση του πολιτικού διαλόγου θα γίνει στις 23 Μαΐου. Και τώρα περνάμε στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2017. Και είναι μεγάλη μας χαρά να καλωσορίζουμε σήμερα τον Αντιπρόεδρο Βίτορ Κωνστάντσου δεν είναι μια κλασική παρουσίαση της ε, επίσης έκθεσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά είναι μια όλος ιδιαίτερη συνεδρίαση σήμερα, καθώς η θητεία του Αντιπρόεδρου Κωνστάνσιο λύγει στις 21 Μαΐου φέτος. Οπότε είναι η τελευταία του παρουσία εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, όχι απλώς μόνο μετά από μία οκταετία, ε, στην ε, στο αξιωμά ως Αντιπροέδρου, αλλά 18 στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αποτείω λοιπόν φοροτιμής στον ρόλο σας και την συνεισφορά σας στις καθοριστικές σημασίες δράσεις που έχει αναλάβει σε αυτό το διάστημα για την Ευρωζώνη η ΕΚΤ, διαφυλάσσοντας την ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα και αυτήν των τιμών και φυσικά όχι μόνο τη σταθερότητα των τιμών, καθώς η ΕΚΤ είχε αποφασιστικό ρόλο και εσείς βεβαίως προσωπικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν, χαιρετίζω την ε, συνεισφορά σας στο κοινό μας έργο και σας εύχομαι καλή τύχη για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε Αντιπρόεδρε Κωνστάξιο. Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ, όπως ξέρετε, έχει δημοσιευθεί στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. και καλύπτει τη χρηματοοικονομική πολιτική, τις ε, οικονομικές εξελίξεις, ε, τι γίνεται με το Euro το, ευρώ, το σύστημα του ευρώ στις διάφορες περιοχές αρμοδιότητα της ΕΚΤΑ, καθώς και την αποστολή της έκθεσης ε, από τον κύριο Ντράγκη προς τον κύριο Ταγιάννη με ένα παράρτημα της ΕΚΤ όπου υπάρχουν απαντήσεις στις ερωτήσεις της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας του 2016 με ε, τότε εισηγητή τον κύριο Χώνας Φερνάντες. Ε, οι απαντήσεις αυτές θα διατεθούν ε, στα μέλη του Κοινοβουλίου ε, και ε, ήδη είναι διαθέσιμα όλα αυτά από τις 3 ε, σήμερα το μεσημέρι. Οπότε θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Κωνστάνσιο. Ξέρετε πώς οργανώνεται αυτή η συζήτηση με χρονοθυρίδες πεντάλεπτες. Αντιπρόεδρο Κωνστάνσιο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας ε, εισαγωγικά λόγια. Σας ευχαριστώ επίσης και για τις ευχές σας όταν ε, θα έχω φύγει από την ε, θέση αυτή. Επιτρέψτε μου να σας πω επίσης ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ για τελευταία φορά στην Επιτροπή σας για να σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για το 2017 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ. Και προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ευρωβουλευτές, τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το καρποφόρο διάλογο που είχαμε μεταξύ μας όλα αυτά τα 8 χρόνια. Έχει αλλάξει πολύ ο κόσμο ε, όλο αυτό το διάστημα. Το ίδιο ισχύει και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οι τιμέ, κυρίω η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε του κινδύνου πολύ χαμηλού πληθωρισμού ή και αποπληθωρισμού μάλιστα, απέτησαν από εμά να διαβρύνουμε την εργαλειοθήκη μα ε, για την ε, αντιμετώπιση τη νομισματική μα πολιτική. Χωρί λοιπόν τι πολιτικέ αυτέ, στα πλαίσια τη νομική μα εντολή, η νομισματική ένωση μπορεί και να έχει καταρρεύσει. Ω λοιπόν συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο για 18 χρόνια, 8 ως αντιπρόεδρος, είμαι περήφανος που μπορώ να πω ότι συνεισέφερα σε αυτές τις πολιτικές. Όμως θέλω να σας υπενθυμίσω ότι οι διάφορες θεσμικές μεταρρυθμίσεις ή έκτακτες που προσθέθηκαν στον μινιμαλιστικό αρχικά σχεδιασμό της Νομισματικής Ένωσης δεν έχουν ολοκληρωθεί και συνεπώς παραμένουν υπαρξιακοί κίνδυνοι ως νομοθέτες ε, και εσείς έχετε συνεισφέρει στις μεταρρυθμίσεις αυτές και ελπίζω, είμαι σίγουρος, ότι θα συνεχίσετε να κάνετε ό,τι είναι αναγκαίο προκειμένου να συμπληρώσετε την ε, Οικονομική Ένωση. Όλα αυτά τα χρόνια έχετε αναθέσει στην έκτη επιπλέον αρμοδιότητες. Ο δικός σας ρόλος είναι να απαιτείται από εμά λογοδοσία και αυτό φαίνεται στις εξελίξεις και ο διάλογος αυτός μαζί σας θα παραμείνει προτεραιότητα για την ΕΚΤ. Είναι μια σταθερή πρακτική που έχουμε πρώτα απ' όλα να προσφέρουμε γραπτό feedback, αντίδραση δηλαδή στη δικιά σας έκθεση μετά από την παρουσίαση της ετήσιας μας έκθεση και αυτό το feedback να ξέρετε ότι σήμερα δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα μας. Στις παρατηρήσεις μου λοιπόν θα συζητήσω για τις επιπτώσεις των αποφάσεών μας όσον αφορά την οικονομία για το 2017 και στη συνέχεια θα αναφερθώ και το σημαντικό ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα για την μετάδοση της νομισματικής μας πολιτικής και πώς μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη. Το 2017 λοιπόν η ανάπτυξη, <clears throat> η οικονομική, ήταν ισχυρή και διευρύνθηκε. Όμως από την άλλη μεριά περιμένουμε ε, σιγά σιγά άνοδο του πληθωρισμού ο οποίος ε, είχε μείνει σε ελεγχόμενα επίπεδα το τελευταίο αυτό διάστημα. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή, προκειμένου να σχεδιάσουμε την πορεία της νομισματικής μας πολιτικής, ε, σταθμίζοντας όλα μας τα μέτρα. Πρέπει να τα επανασταθμίσουμε ακριβώς, λαμβάνοντας υπόψη τι νομισματικά κριτήρια χρειάζονται και να δούμε πώς θα φτάσουμε τον πληθωρισμό στα επίπεδα που θέλουμε. Στις αρχές του 2017 η ανάκαμψη της οικονομίας στην Ευρωζώνη ήταν σταθερή. Όμως ο κίνδυνοι παρέμεναν προκειμένου να πάνε τα πράγματα προς τα κάτω. Στα μέσα της χρονιάς η ανάπτυξη ενισχύθηκε περισσότερο και υπήρχε μεγαλύτερη επέκταση και πιο γρήγορα από ό,τι περιμέναμε νωρίτερα οι πιθανότητες να έχουμε ένα κακό σενάριο, όπως για παράδειγμα οι αποπληθωριστικοί κίνδυνοι, εξαφανίστηκαν από το τοπίο. Και γι' αυτό προσαρμόσαμε τις κατευθυντήριες γραμμές μας και αφαιρέσαμε την μία σε επιπλέον ε, περικοπές στα επιτόκια. Στη συνέχεια μέσα στην χρονιά είχαμε και τη διασφάλιση ότι ο πληθωρισμός σιγά σιγά ε, σύγκλινε προς το στόχο μας. Παρ' αυτά, οι εξελίξεις των ε, τιμών ε, συνέχιζαν υπό έλεγχο και μέτρα για το βασικό πληθωρισμό έδειχναν ε, μια τάση προς τα πάνω. Και αυτό ήταν το πλαίσιο λοιπόν, μέσα στο οποίο πήραμε τις αποφάσεις μας τον Οκτώβριο. Πιο συγκεκριμένα ανακοινώσαμε τότε ότι θα μειώναμε την ένταση της αγοράς κεφαλαίων μηνιαία στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Συγχρόνως επεκτείναμε και τον ορίζοντα για την αγορά των κεφαλαίων μέχρι στα τέλη του Σεπτεμβρίου του 2018 ή και ακόμα πιο πέρα αν αυτό είναι αναγκαίο και όπως και να έχει το πράγμα μέχρι το Διοικητικό Συμβούλιο να δει ότι έχουμε φτάσει όσον αφορά τον πληθωρισμό πολύ κοντά στους στόχους μας. Επιπλέον αποφασίσαμε να επεκτείνουμε και τις ε, διαδικασίες ε, ε, προσφοράς ε, τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2019 και να παρακολουθήσουμε και να, ε, παρετέρω την κατάσταση όσον αφορά τον πληθωρισμό. Μέσα στο 2017 τα νομισματικά μας μέτρα συνέχισαν να στηρίζουν δανειστικές συνθήκες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενισχύοντας την ε, ροή ρευστού σε όλη την Ευρωζώνη. Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα τα οποία χρειάστηκαν από τα μέσα του 2014 και αυτά που αποφασίστηκαν τον Οκτώβριο του 2017, οι συνολικές επιπτώσεις στο πραγματική αύξηση ΑΕΠ και τον πληθωρισμό μέσα στην ε, Ευρωζώνη φαίνεται να είναι 1,9 ε, μονάδες ποσοστιαίας συσσωρευτικά για την περίοδο ανάμεσα στο 2016 και το 2020. Επιτρέψτε μου τώρα να επιστρέψω στο ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα στην μετάδοση της νομισματικής μας πολιτικής. Η βασική δομή του μη χρηματοπιστωτικού τομέα άλλαξε πάρα πολύ τα τελευταία 10 χρόνια παίζει πλέον πολύ σημαντικό ρόλο στην μετάδοση της νομισματικής μας πολιτικής προς την πραγματική οικονομία και βοηθάει την αντοχή μας σε σοκς. Ε, αντίθετα με ό,τι έγινε στις Ηνωμένε Πολιτείε, στη δικιά μας την περίπτωση παραδοσιακά το τομέας αυτός βασίζεται κυρίως στις τράπεζες για να χρηματοδοτηθεί. Όμως αυτό άλλαξε δραστικά γιατί οι μη τραπεζικές ε, οικονομικές πηγές ε, φάνηκε να είναι πιο σημαντικές ε, μετά την οικονομική κρίση. Τα συνολικά κεφάλαια επενδυτικών κονδυλίων ποσοστία και στα κεφάλαια των τραπεζών πήγαν από 16% το 2007 στο 44% πέρυσι. Και τα δάνεια τώρα, ποσοστία των τραπεζών στο συνολικό απόθεμα των ε, επιχειρήσεων εκτός χρηματοδότης μέσα στο 2017 ήταν μόλις πάνω από 12%. Και λαμβάνοντα υπόψη μόνο τα μέσα χρέους, equities κλπ, το ποσοστό των ε, τραπεζικών δανείων στο σύνολο του χρέους αυτού ήταν μόνο 28% πέρυσι. Η νομισματική πολιτική και τα σχετικά μέτρα που ελήφθησαν από τα μέσα του 2014 είχαν σημαντικές επιπτώσεις στην ε, μετάδοση αυτή. Οι εκτιμήσεις μας λένε ότι η αύξηση των ε, δανείων θα ήταν ε, η μισή χωρίς τα δικά μας μέτρα. Ουσιαστικά ενισχύσαμε τους ισολογισμούς, την ισορροπία στους ισολογισμούς, δηλαδή με τα μέτρα αυτά βασιζόμενοι στα ομόλογα. Επιπλέον τα μέτρα μας αύξησαν και το μερίδιο των μη τραπεζικών οικονομικών πηγών στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη. Το πρόγραμμα αυτό ενθάρρυνε την έκδοση ομολόγων και μείωσε την απόδοση. Κάτι το οποίο βοήθησε και τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πολύ βασικό για περισσότερες επενδύσεις και για μεγαλύτερη διαφοροποίηση πηγών χρηματοδότησης όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Κάτι το οποίο ενισχύει την αντοχή. Και έτσι απελευθερώθηκε πεδίο στον ισολογισμό των τραπεζών ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τις πιστώσεις τους προς τις μικρότερες εταιρείες. Το δεύτερο θέμα είναι ότι η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ μπορεί να ωφεληθεί από ένα σταθερό χρηματοοικονομικό τομέα. Γι' αυτό ήθελα να στραφώ στους κινδύνους και τις πολιτικές ε, μακροπροληπτικού χαρακτήρα στην Ευρωζώνη και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις που χρειάστηκαν σε νομοθετικό επίπεδο. Η χρηματοοικονομική σταθερότητα του, της Ευρωζώνης εξελίχθηκε θετικά το 2017 με καλές οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, τέσσερις βασικοί κίνδυνοι παρέμειναν και πρέπει να ελέγχουν ελέγχονται ακόμη. Πρώτα απ' όλα, ο κίνδυνος μιας ε, αντιστροφής στα premium των κινδύνων διεθνώς στις χρηματοοικονομικές αγορές είναι κάτι που θα πρέπει να συνεχίσουμε να διερευνούμε και το 2017 για να δούμε τι αποδόσεις θα έχουν. Δεύτερον, οι τράπεζες της Ευρωζώνης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κερδοφορίας σε σχέση με τις, ε, με τις δυσκολίες ως προς το κόστος ε, και το αποθεματικό τους σε μακρύς Διάρκεια δάνεια. Τρίτον, υπάρχουν υψηλά επίπεδα χρέου και για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, χωρί να μπορούν να αποπληρωθούν με βεβαιότητα. Και τρίτον, υπάρχει και το πρόβλημα τη αναντιστοιχία στι ρευστότητε και τη ελληπού ανάπτυξη του επενδυτικού τομέα. Υπάρχουν και κίνδυνοι στον ε, μεσητικό τομέα, τον τομέα των ακινήτων. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σχεδιάσουμε αναλόγω τι μακροπρόληπτικέ μα ε, πολιτικέ. Υπήρξαν αναντιστοιχίες στην Ευρωζώνη, ιδίως στην αγορά των ακινήτων συνολικά, ενώ αυξήσεις των τιμών σε κάποιες χώρες ε, απέτησαν σωστή απάντηση με ανάλογα μέτρα μακροπροληπτικών πολιτικών. Η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των επιμέρους μέτρων δείχνει ότι υπάρχει μια ανάγκη ανάμειξης διαφορετικών εργαλείων με ευρύτερα μέτρα όπως τον περιορισμό των ε, δανείων που δίνονται βάσει της αξίας ή των ε, χρεών που αναλαμβάνονται και του λόγου μεταξύ τους ώστε να ελεγχθεί η έκθεση και οι κεφαλαιακές απαιτήσει. Επίσης, ε, τα εργαλεία δεν προβλέπονταν στον σχετικό κανονισμό IVCRR. Έτσι λοιπόν χρειάστηκαν τουλάχιστον δύο ε, νέα εργαλεία για να συνδυαστούν αυτά με τις δημόσιες αρχές όπως ε, προέβλεπε το άρθρο 458 του Γενικού Κανονισμού. Αυτό επέτρεψε στις αρχές μακροπροληπτικής φυσίωση να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα ο έγκαιρος εντοπισμός των συστημικών κινδύνων και της ανάληψης τέτοιων μέτρων ήταν κάτι που μας επέτρεψε να ε, έχουμε χρηματοοικονομική σταθερότητα με τον ανάλογο χρηματοοικονομικό κανονισμό. Ήταν ο μόνος τρόπος ε, από την κρίση και μετά. Όλοι οι σχετικοί κανόνες του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματος έχουν ε, μεταρρυθμιστεί και αποπερατωθεί στο πλαίσιο της Βασιλείας 3. Βέβαια το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να ε, αναζητήσουμε τους στόχους της Τραπεζικής Ένωσης για να βελτιώσουμε τη σταθερότητα του σημείου. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει ένα καθοριστικό ρόλο για να δραματίσει εδώ. Η μείωση του κινδύνου έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ε, λόγοι των ε, ε, μάλλον τα κεφάλαια των τραπεζών βρίσκονται σε καλά επίπεδα, ενώ εφαρμόζεται ο κανονισμός MRAL και όπως προβλέπεται και στο σχετικό κανονισμό BRD θα πρέπει να υπάρξει ενδεχομένως παρέμβαση του Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας για τον έλεγχο του χρέου και τη σχετική μόχλευση. Θα πρέπει όμω να αναλάβουμε δράσεις σε τρει τομεί. Πρώτα απ' όλα να εναρμονίσουμε και να βελτιώσουμε το πλαίσιο αφαιρεγγιότητα. Δεύτερον, να έχουμε συστηματικέ αναθεωρήσει ε, και ελέγχου για το τι γίνεται με τα δάνεια που δεν αποπληρώνονται. Τρίτον, να δούμε ποιε είναι οι εθνικές, ε, ε, το εθνικό πεδίο διακριτικής ευχέρεια, ώστε η ΕΚΤ να εφαρμόσει σωστά την εποπτεία του τραπεζικού συστήματο τη Ευρωζώνη. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ε, πρέπει να δει τη φεραγγιότητα και το backstop για τη ρευστότητα σε επίπεδο ενό κοινού ταμείου. Αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το πετύχουμε για να βελτιώσουμε την συνολική εξοπιστία του μηχανισμού μηχανισμού ε, διάσωσης. Ε, τώρα, ω τον, ε, εκτός τον εξωτραπεζικό τομέα, είναι σημαντικό η προληπτική πολιτική μα να εφαρμοστεί στα πλαίσια τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη πραγματική οικονομία. Η αυτή την έννοια, καλωσορίζω την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στηρίξει τι μεγάλε επενδυτικέ εταιρείε με δραστηριότητε που θα μπορούσαν να τι ταυτίζουν με, τους χρηματοπιστωτικούς, με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και αυτό να τι εντάσσει στο σύστημα υποπτία. Βεβαίω, θα πρέπει να φροντίσουμε η νομισματική μας πολιτική να έχει τέτοιου κανόνες που να αντιμετωπιστεί η αστάθεια αλλά να βελτιωθεί και να, να υπάρξει και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Είδαμε περιορισμό στην παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού από, το, από τη δεκαετία του 1990 και μείωση κατά 1% σε δυνατότητες ανάπτυξης συνολικά. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε αυτό και να δούμε τη διαφορά μεταξύ των πρωτοπόρων και των ε, τελευταίων των οραγών εταιριών με την σωστή απόδοση των κεφαλαίων. Θα πρέπει να είναι υγιής ο τραπεζικός τομέας με εύρυθμος, με σε λειτουργούσες τραπεζικές και κεφαλαιοχικές αγορές ώστε να βελτιωθεί η ανάπτυξη. Η ΕΚΤ έχει στηρίξει τις αγορές κεφαλαίων ως τώρα ε, διαφοροποιώντας τις πηγές χρηματοδότησης για μη χρηματοδοτικές εταιρείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της νομισματικής πολιτικής. Αλλά και η Ένωση Κεφαλαίων Αγορών είναι σημαντικό για να ε, απεπερατωθεί η Τραπεζική Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν καλώ όλους τους ενδιαφερομένους να, τον, να τονώσουν τις προσπάθειές τους για να πετύχουμε αυτή την Ένωση Κεφαλαίου αγορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας ολοκληρώσω. Ένα από τα βασικά διδάγματα της κρίσης για την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ είναι ότι με τα μέτρα μας και τις πολιτικές μας πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες του τραπεζικού ε, τομέα όπου υπάρχουν. Και ενώ είναι σημαντικό να παρακολουθούμε τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ε, ε, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει η εφαρμογή των μέτρων από τους σωστούς διάβλους. Θα πρέπει να ε, επιτελεστεί περαιτέρω πρόοδος για την Τραπεζική και Ένωση και την Ένωση των Κεφαλαίων Υπ' αυτήν την έννοια πιστεύω ότι με την πολύ καλή επικοινωνία που έχουμε μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και ΕΚΤ θα καταφέρουμε και μετά την οκταετή μου εμπειρία να διαδραματίζουμε εδώ ένα σημαντικό και θετικό ρόλο στην ολοκλήρωση αυτών των προσπαθειών. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ο πρόεδρο Γκαλθιέρη, σα ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε για τα στοιχεία που παραθέσατε και βεβαίως και το Κοινοβούλιο δεσμεύεται στους φιλόδοξους αλλά αναγκαίους αυτούς νομοθετικούς στόχους στους οποίους παραπέμψατε στην ομιλία σας. Και θα συνεχίσουμε βεβαίως την καρποφόρο διαθεσμική συνεργασία ε, μεταξύ ημών Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης δηλαδή και ημών δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με ανταλλαγή επιστολών και βεβαίως για, για τον διορισμό του διαδόχου σας. Θα αρχίσουμε εδώ τι παρεμβάσει. Πρώτος ο κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης για τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας εκφράζω τις ευχαριστίες μου προσωπικά αλλά και της πολιτικής μου ομάδας για την επικοδομητική συνεργασία που είχαμε μαζί σας τα τελευταία 8 χρόνια. Έχουμε την δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του έτους 2017, την οποία αναμέναμε με μεγάλη ανυπομονησία. Την προηγούμενη χρονιά εσείς και οι συναδελφοί σας, για πρώτη φορά από την οικονομική κρίση του 2008, δείχνεται μια προσεκτική αλλαγή κατεύθυνση στην ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική να, και έχετε αρχίσει την μείωση, τη σταδιακή μείωση των ε, αγορών χρήματος, των, ε, της ε, ποσοτικής χαλάρωσης, διότι το μακροοικονομικό πεδίο αναπτύσσεται και μάλιστα όχι από την αρχή του τρέχοντος έτους, θετικά σε ολόκληρο Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ένα μέσο όρο πληθωρισμού 1,4%. Η οικονομική ανάπτυξη σημειώνεται ήδη θετικά από την αρχή του 2017. Παρ' όλα αυτά, εσείς προτείνετε μια αργή αλλαγή στην νομισματική πολιτική, ενώ η Αμερικανική Fed, για παράδειγμα, προβλέπει σημαντική μείωση του δικού της ισολογισμού, του δικού της balance sheet, από τη δική σας τράπεζα ακούμε μόνο πολύ προσεκτικές τοποθετήσεις. Γι' αυτό και σας ρωτώ σήμερα, ποιες είναι οι προσδοκίες σας σε ό,τι αφορά την μακροπρόθεσμη εξέλιξη του ισολογισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δεύτερο, εάν ο ισολογισμός, αυτό το balance sheet, θα παραμείνει τόσο, θα το πω καθαρά παραφουσκωμένο, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ενδεχομένως συνεπάγεται αυτή η εξέλιξη. απάντηση του κυρίου Κωνστάνσιου. Σας ευχαριστώ πρώτα για τα καλά σας λόγια. Ε, τώρα για την ερώτησή σας. Ναι, υπήρξαμε προσεκτικοί και ιδίω σε σύγκριση με τις εξελίξεις στις Ηνωμένε Πολιτείε. Όμως οι οικονομικοί κύκλοι στις δύο αυτές περιοχές του κόσμου κινούνται διαφορετικά. Ο πληθωρισμός που είναι ο δικός μας αντικειμενικός στόχος δεν έχει ανταποκριθεί ακόμη απολύτως στα, στις προσδοκίες μας μιλήσατε για το ρυθμό του 1,4 του Μαρτίου. Τον Φεβρουάριο όμως ήταν 1,1 μόνο. Εξάλλου, όπως βλέπετε και όπως γνωρίζετε, στα τελευταία σχεδόν τέσσερα χρόνια ο εγχώριος πληθωρισμός είχε μείνει στο 1 περίπου της 100. Το να αναμένει λοιπόν κανείς μια μελλοντική εξομάλυνση των ε, ρυθμών του πληθωρισμού ε, είναι υπεραισιόδοξο. Είδαμε τον Οκτώβριο όμως ότι εμείς είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε την πολιτική μας ε, ανάλογα με τις εξελίξεις. Και είμαι βέβαιος ότι η πορεία αυτή θα ε, ακολουθηθεί και στο μέλλον, καθώς θα βελτιώνεται η κατάσταση, ελπίζω. Και πράγματι έχουμε την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να εξελίσσεται παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις που κάνουμε, το κάνει το προσωπικό μας, τα projections, προβλέπουν για φέτος 1,4 και πάλι για του χρόνου 1,4. Άρα η διαδικασία είναι όντως πολύ σταδιακή και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να αποφύγουμε κάποιες ε, έντονα περιοριστικές πολιτικές να ε, οδηγήσουν ε, σε λάθος κατεύθυνση. Νομίζω λοιπόν ότι η πολιτική μας αποδίδει. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα έκτακτα μέτρα τα οποία έχουμε υιοθετήσει κάποια στιγμή θα λήξουν και μετά θα ακολουθήσει μια διαδικασία μείωσης του ισολογισμού της ε, Κεντρικής Τράπεζας. Παρ' όλα αυτά, βεβαίως δεν ξέρω, δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα φέρει το ε, μέλλον και ούτε θα μπορώ πλέον να το επηρεάσω. Αλλά τονίζω ότι στις ΗΠΑ προηγήθηκε μακρά συζήτηση σχετικά με το μέλλον του ε, ισολογισμού της Κεντρικής Τραπεζάς τους και δεν είναι ακόμη καθαρό εάν η Fed επανέρχεται στον ίδιο τύπο balance sheet όπως πριν από την κρίση ή αν θα παραμείνει, όχι βέβαια στα ίδια επίπεδα, θα υπάρξει μια σημαντική μείωση, αλλά αν θα διατηρήσει κάποιο σημαντικό μέγεθος στο balance sheet. Και υπάρχουν λόγοι που έχουν σχέση και με την ε, νομισματική σταθερότητα, αλλά και με το γεγονός επίσης ότι συνολικά σε ολόκληρο τον κόσμο και όπως είπα και στην τοποθέτησή μου και στην Ευρώπη, οι τράπεζες περιορίζουν το ρόλο τους στη χρηματοδότηση των οικονομιών. Το δίκτυο λοιπόν επιτοκίων που θα επηρεάζεται από την νομισματική πολιτική γίνεται πλέον περίπλοκο, διότι δεν περνάμε μόνο μέσα από τις τράπεζες. Και αυτό είναι και ένα από του λόγου που κρύβονται πίσω από αυτή τη συζήτηση που γίνεται στι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι ένα απλό σχόλιο που κάνω. Προ Θεού δεν κρύβεται από πίσω καμία πρόθεση άσκηση πολιτική. Είμαι βέβαιο ότι θα μειώσουν, θα μειωθούν όλοι οι ισολογισμοί των κεντρικών τραπεζών που χρειάστηκε και εδώ και στι Ηνωμένες Πολιτείες και στον Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιαπωνία να λάβουν αυτά τα έκτακτα μέτρα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εγώ. Να συνεχίσουμε με αυτό που είπε ο κύριος Μπάλτς, αλλά από μια διαφορετική σκοπιά. Λέτε στην έκθεσή σας ότι η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει να είναι σόφρον. Αυτό σημαίνει να επανέλθει ε, σε μια ομαλή κατάσταση διότι οι εξελίξεις των τιμών, όπως θυμήσατε, εξακολουθούν να είναι οι εξελίξεις δηλαδή πάρα πολύ περιορισμένες. Τα έχουμε συζητήσει αυτά και τα έχουμε συζητήσει και με τον ίδιο τον πρόεδρο Ντράγκη. Και είπε ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους ε, όσο και η δυναμική της αύξησης των μισθών παραμένει πάρα πολύ περιορισμένη. Πάντως, ξεκινώντας από αυτό, μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στην ετήσια εκθεσή σας Βάζετε δύο θέματα, το ένα μετά το άλλο. Πρώτο, στη σελίδα 22. Μιλείτε για διαρθρωτικέ μεταρρυθμίσεις που λέτε ότι αυτές συνέβαλαν στην αύξηση της απασχόλησης. Και μετά αναφέρεστε σε μια business survey για να δείξετε ποια θα είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση που πρέπει να συνεχιστεί. Περαιτέρω ευκαμψία στην αγορά εργασία προσπάθεια να γίνουν οι σχετικέ. Ε, συνθήκες πιο εύκαμπτες και να χαλαρώσει και η προστασία της ανεργίας. Αυτά βλέπουμε που λέτε εδώ. Και μετά πηγαίνουμε στο επόμενο κεφάλαιο της, ε, ε, της έκθεσης. Ποια είναι, γιατί δεν λειτουργεί η καμπύλη Φίλιπς και στην έκθεση εντοπίζει γιατί η καμπύλη Φίλιπς δεν αποδίδει τόσο καλά. Και ίσως εν τέλει, λέτε, υπάρχει μια μεταρρύθμιση που πρέπει να γίνει και στι συλλογικέ συμβάσει, δηλαδή στη διαδικασία συλλογικών συμβάσεων. Εγώ τα βρίσκω αυτά λίγο αντιφατικά. Δηλαδή, από τη μια μεριά προτείνεται μια ατζέντα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε συνέχεια ε, των κλασικών αντιλήψεων. Από την άλλη μεριά όμως αναγνωρίζεται ότι είναι και ένα από τα προβλήματα που ε, μάλλον ένας από τους λόγους που έχουν μειώσει τον τόνο, την ε, δυναμική της αύξησης ε, μισθών αλλά και παραγωγικότητας κλπ. Βέβαια, οι επιχειρηματίε μπορεί να θεωρούν ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά πράγματα. Υπάρχουν όμω και άλλε απόψει που μπορούν να διοχετευτούν ω συμβουλέ στο έργο τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστώ, απαντά ο κ. Κωνσταντζιο. Όπω ε, υπενθυμίσατε, η έκθεση από την οποία αναφέρατε δεν είναι παρά ε, ένα συμπίλημα απόψεων ε, επιχειρήσεων που έχουν απαντήσει στην έρευνα σε business survey. Είναι λοιπόν η δική του γνώμη, την οποία, την ζητήσαμε για να δούμε. Το λέω αυτό για να τονίσω ότι πράγματι δέχεται να υπάρχουν αντιφάσεις και αυτό ίσως είναι και αναμενόμενο. Διότι τέτοιου είδου αλλαγέ θέλουν να δουν βέβαια οι διοικητέ των επιχειρήσεων, οι μάνατζερ. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι και η μεγάλη συζήτηση που γίνεται στι κοινωνίε μα για τα προβλήματα αυτά. Και η κατάσταση σε ό,τι αφορά την ευκαμψία τη εργατική νομοθεσία συνολικότερα είναι πολύ διαφορετική μέσα στη ζώνη ευρώ. Δεν υπάρχει κανένα ιδιαίτερο benchmark. Και αν ακόμα πάρετε τις πιο ανεπτυγμένες και ισχυρότερες οικονομικά χώρες, θα δείτε για παράδειγμα στη δημοσίευση του ΟΣΑ των δικτών της ευκαμψίας ε, της αγοράς εργασίας, η χώρα που έχει τη χαμηλότερη ευκαμψία στην εργατική νομοθεσία είναι η Γερμανία. Διότι το σύνολο μεταρρυθμίσεων που έγιναν σε πολλές χώρες στη διάρκεια της κρίσης άλλαξε το τοπίο, άλλαξε το πανόραμα με πολύ σημαντικό τρόπο και μπορεί να δει κανείς ότι μέρος της ανάκαμψης η οποία ακολούθησε αργότερα με κάποια χρονική υστέρηση μετά από τις μεταρρυθμίσεις και επομένω και η αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μπορούν όντως να αποδοθούν στις μεταρρυθμίσεις αυτές. Είναι γνωστό επίσης και υπάρχουν και εμπειρικά αλλά και, και εμπειρικές και πανεπιστημιακές ε, ε, μελέτες που δείχνουν ότι οι διαφορετικές μεταρρυθμίσεις όταν αναφέρονται Στι μεταρρυθμίσει ε, στο πλαίσιο της αγοράς εργασία, οι μεταρρυθμίσει αυτές συνήθως έχουν ένα αρχικό αποτέλεσμα μείωση του επίπεδου των αμοιβών. Αυτό είναι γνωστό, είναι πασίγνωστο. Και γι' αυτό πράγματι γίνεται η παραπομπή όταν συζητεί κανείς την σχέση της καμπύλης Φίλιπς, του βαθμού δηλαδή της ανεργίας και της απόδοσης του πληθωρισμού ότι πράγματι υπάρχει μια περίοδος εντατικ... όταν υπάρχει μια περίοδος εντατικών μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια της αγοράς εργασίας αυτό οδηγεί σε μείωση των αμοιβών, υπερομισθείων Η ανταπόκριση λοιπόν σε αυτή την περίοδο αμέσως μετά την μεταρρύθμιση μειώνει και την ανταπόκριση του πληθωρισμού στις ε, συνθήκες τη αγορά εργασία. Δεν πρόκειται για αντίφαση, είναι ζήτημα χρονισμού. Γουαλτιέρι. Ναι, βέβαια, το, δεύτερο, θέμα είναι καλά η πρώτη φορά, αλλά τι γίνεται τη δεύτερη φορά. Θα πρέπει να αφιστούν τότε. Κωνστάνσιο, υπάρχει και κάτι άλλο. Είναι σημαντικό επίση, διότι δείχνει πολλέ από τι δημοσιεύσει και μελέτε που έχουμε κάνει και μια μεγάλη μελέτη για τον πληθωρισμό και την απόδοση του πληθωρισμού που δημοσιεύσαμε, το λεγόμενο Lift Project, το βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας αυτό, όπου βλέπετε ότι αντιθέτως από τις ΗΠΑ και αλλού, η καμπύλη Phillips, δηλαδή ο βαθμός ανταπόκρισης του πληθωρισμού στη μείωση απόδοσης της οικονομίας, αυξάνεται τελευταία. Και αντίθετα λοιπόν από τις ΗΠΑ, η αύξηση της καμπύλης, η, ε, αν, αν α ας πούμε της καπήλης είναι σημαντικότερη. Και αυτό είναι γνωστό στους οικονομολόγους. Ότι αυτό είναι το αρχικό αποτέλεσμα των διαρθωτικών μεταρρυθμίσεων και μετά, ως αναμενόταν βεβαίως, αυξάνεται η κάμψη της καμπύλης. Μπέντ Λούκε. Καλημέρα κύριε Κωνστάνσιο, θα μιλήσω γερμανικά. Ερώτηση για την ε, σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίω των τραπεζών στην Ευρωζώνη και πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία. Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρεται στην εκθεσή της στην κατάσταση αυτή, αλλά με λίγα λόγια. Εντοπίζεται κατά βάση δύο παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών. Μιλείτε για τα χαμηλά επιτόκια και μιλείτε και για τη χαμηλή απόδοση των καταθέσεων. Δεν αναφέρεστε όμως στον πολύ χαμηλό πληθωρισμό που καθιστά τις παραδοσιακές κλασικές ε, επιχειρήσεις δράσης των τραπεζών, δηλαδή την χορήγηση πιστώσεων, στην πραγματικότητα μη κερδοφόρα. Και αυτό οδηγεί ώστε οι τράπεζες να πιέζονται να ασκήσουν περισσότερο investment banking, δηλαδή να επενδύουν. Και εν ώψη μάλιστα και της κρίσης στην Deutsche Bank που πάλι εμφανίζεται στους ε, τίτλους των εφημεριδών ασφαλώς και δεν πρόκειται να σχολιάσετε την περίπτωση του Deutsche Bank, το γνωρίζω αυτό. Πρόκειται όμως για ένα σημαντικό πρόβλημα. Αντιμετωπίζει και αυτή μια παρόμοια κατάσταση και η Commerzbank στη Γερμανία επίσης. Ερωτώ λοιπόν, ποια ευθύνη φέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την μη ικανοποιητική ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων σημαντικών τραπεζών που πρώτα-πρώτα φάνηκε να περνούν αυρόχης ποσή από την κρίση, τώρα όμως εκ των υστέρων εν ώψη της εξελίξεως των επιτοκίων αντιμετωπίζουν βαρύτατες δυσχέρειες για να ασκήσουν τις κλασικές παραδοσιακές δραστηριότητες με κερδοφόρο τρόπο και θεωρείται ότι μπορεί να αλλάξει πολιτική η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε να καταστήσει κερδοφόρα την, την τραπεζική δραστηριότητα και στη Γερμανία αλλά και στις άλλες χώρες της ζώνης ευρώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Πρώτα απ' όλα, το θέμα της κερδοφορίας των τραπεζών μεταξύ χωρών αλλά και μέσα στην ίδια χώρα ε, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν είναι τόσο ο χαμηλός πληθωρισμός που εξηγεί τις διαφορές της κερδοφορίας. Αυτό ισχύει μέσα στην Ευρωζώνη, αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα εκτός Ευρωζώνης. Σουηδία. Εκεί τα επιτόκια είναι χαμηλότερα από ό,τι αυτά που έχουμε εμείς στην Ευρωζώνη. Χαμηλότερα. Έχουν αρνητικά 0,75, κάτι τέτοιο. Οπότε, παρόλα αυτά, οι τράπεζές τους εκεί έχουν απόδοση 12% σχεδόν. Στην περίπτωση της Ευρωζώνης, με τις 16 σημαντικές τράπεζες, στο τρίτο τρίμηνο είχαμε μια απόδοση 7% κατά μεσόρο. Ενώ εκεί είναι 12%. Όταν λοιπόν κοιτάξει κανείς, συγκρίνει και προσπαθήσει να καταλάβει γιατί, η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι πρόκειται για την διαφορά κόστους και αποτελεσματικότητας των τραπεζών. Αν υπολογίσετε το λόγο συνολικού κόστους των τραπεζών και συνολικού ενεργητικού, κόστος και ενεργητικό, τότε η αναλογία αυτή, ο λόγος αυτός στις βόρειες τράπεζες, στη Σουηδία κυρίως, είναι το μισό από ό,τι έχουμε στην Ευρωζώνη. Το μισό. Και είναι και πιο ψηλό στη Γερμανία από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αν ε, κοιτάξετε μάλιστα στην ιστορία, ο μέσος όρος κερδοφορίας των γερμανικών τραπεζών ήταν χαμηλότερος από ότι γενικά στην Ευρώπη για λόγους εντάξει κατανοητούς που δεν είναι της παρούσης και δεν έχουν να κάνουν με κάποια αρνητική αντιμετώπιση. Υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι γι' αυτό. Πάντως αυτό το λέω για να σας δείξω ότι το εύρος κερδοφορίας των τραπεζών και οι διαφορές που βρίσκουμε μεταξύ χωρών αλλά και μέσα στην ίδια τη Γερμανία μόνο δεν εξηγείται μόνο από τα χαμηλά, το χαμηλό, τα χαμηλά επιτόκια. Μα δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου, λέει ο κ. Λούκα. Θα έρθω, θα έρθω. Περιμένετε, κάνω πρώτα αυτές τις ε, παρατηρήσεις για να σας δώσω το πλαίσιο, γιατί η ερώτησή σας μου έδωσε την εντύπωση ότι υπονοείται πως φταίνε τα χαμηλά επιτόκια για την χαμηλή κερδοφορία. Και όπως ακριβώς σας εξήγησα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα μέσα στην Ευρωζώνη και εκτός Ευρωζώνης που δείχνουν ότι δεν ισχύει αυτό. Έχει να κάνει σε μερικές χώρες με τα MPLs, δεν λέω ότι αυτό ισχύει στη Γερμανία, στις γερμανικές τράπεζες, αλλά αν κοιτάξετε αυτή την αναλογία κόστους ενεργητικού, θα δείτε ότι εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη εξήγηση για τις διαφορές. Στις Ηνωμένε Πολιτείες, ε, να ξέρετε ότι ε, έφτασε σε πιο ισόρροπα επίπεδα η γραμμή, το διάγραμμα εκεί πέρυσι. Και παρόλο που η κατάσταση επηρεάστηκε βέβαια από νομισματικά μέτρα και στη δικιά μας την περίπτωση εξακολουθούμε να αγοράζουμε μέσω πρόθεσμα, όχι πια στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντως τα επιτόκια επηρεάζονται περισσότερο από την αντίληψη, από τη συμπεριφορά των επενδυτών σε ομόλογα. Και το γεγονός ότι η καμπύλη πέφτει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει να κάνει ακριβώς με την αντίληψη των επιδητών ότι πρώτον στα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρξει μεγάλη ανάπτυξη, μεγάλος πληθωρισμός και γι' αυτό παραμένουν χαμηλά τα επιτόκια. Οπότε δεν είναι μόνο η νομισματική πολιτική που ευθύνεται για τα σχετικά επίπεδα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα των επιτοκίων. Άρα δεν μπορείτε να αποδώσετε την ε, κατάσταση της καμπύλης αυτής μόνο στην νομισματική πολιτική, αλλά σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο ε, συγκυρίας που οδηγεί τους επενδυτές να επηρεάζουν με αυτό τον τρόπο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ευχαριστούμε, κύριο Βόλφ Κλίντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πρόσφατες εκλογές στην ε, Ιταλία δείχνει ότι τελικά δεν υπάρχει μόνο διαγωνισμό ποιο είναι υπέρ ή κατά της Ευρώπης και επιπλέον φαίνεται ότι τα κόμματα εκεί δεν είναι γνωστά για να θέλουν να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις. Οπότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η δικιά σας η θέση, ποια είναι όσον αφορά την αξιολόγηση αυτών των εξελίξεων. Φοβάστε ότι μπορεί να αποτελέσει μεγάλη απειλή η Ιταλία για την Ευρωζώνη. Δεύτερον, τα νούμερα και εξέλιξη δείχνει ότι πάμε προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω και η γερμανική Bundesbank φτάνει τα 900 δισεκατομμύρια. Σε αντίθεση με τις Ηνωμένε Πολιτείες, όπου τα μέλη του συστήματος Fed εκεί υποχρεώνονται μία φορά το χρόνο κάθε Απρίλιο να κάνουν την αξιολόγηση, αυτό δεν ισχύει στην Ευρωζώνη. Εσείς βλέπετε να υπάρχει καμία δυνατότητα να διορθωθεί αυτό. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι πατέρες της Ευρωζώνης δεν είχαν σκεφτεί τις εξελίξεις που έχουμε σήμερα. Και τρίτη ερώτηση, τι πιστεύετε για την πρόταση Μακρόν, ο οποίος θέλει να εισαγάγει έναν προπολογισμό Ευρωζώνης, 3 με 4% του ΕΠ, σε αυτή τη τάξη, που είναι αρκετά σημαντικό ποσό, θέλει να έχει Υπουργό Οικονομικό στην Ευρωζώνη και ένα Κοινοβούλιο της Ευρωζώνης. Ποια είναι η γνώμη σας. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Πολύ ευρίες. Και δεν ξέρω κατά πόσο είμαι σε θέση να τις απαντήσω όλες. Τέλος πάντων, για την Ιταλία δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. είναι στα χέρια της Ιταλίας και των Ιταλών να προχωρήσουν στις πολιτικές τους επιλογές και εξελίξεις και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Δεν έχω να κάνω προβλέψεις. Για το Target 2. Θα πάρει πολύ χρόνο, έτσι. Περί τίνος πρόκειται. Πρόκειται για έναν αντικατοπτρισμό δεδομένου ότι οθετήσαμε το κοινό νόμισμα. Αυτό που κάνει το Target 2 είναι ότι δείχνει ποιες είναι οι ροές διαφορετικών πηγών συναλλαγών διασυνοριακά μέσα στην Ευρωζώνη και εκφράζεται βέβαια σε ευρώ. Το αποτέλεσμα είναι ότι Δεν πρόκειται για έναν μηχανισμό ο οποίος να προσφέρει πιστώσεις σε οικονομικούς παράγοντες της μιας ή της άλλης χώρας. Μέλος έχουν ευρώ. Και όταν τα ευρώ πρέπει να πληρωθούν εκτός χώρας, τότε περνάνε μέσα από τις τράπεζες και την κεντρική τράπεζα βέβαια για να καταλήξουν στον τελικό προορισμό. Και τι έχουμε στη διάθεσή μας τότε, ευρώ. Και αν για παράδειγμα η οργάνωση του ευρωσυστήματος ήταν διαφορετική και κάθε δραστηριότητα του ευρωσυστήματος ήταν κεντρικά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε δεν θα βλέπατε καθόλου εθνικούς στόχους προς εξισορρόπηση υπήρχε παγίωση στους κεντρικούς ισολογισμούς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι αν μια χώρα έβγαινε από την Νομισματική Ένωση, τότε η Κεντρική Τράπεζα αυτής της χώρας που έχει ευθύνε απέναντι στις άλλες κεντρικές τράπεζες, αυτό θα ίσχυε, αλλά μόνο στην περίπτωση που μια χώρα έβγαινε από την Ευρωζώνη. Όχι αλλιώς. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση σκεφτείτε και ότι όλες οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν θετικό ενεργητικό. Το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο από το παθητικό. Οπότε έχουν την ικανότητα αυτή να προβούν σε πληρωμές εφόσον χρειαζόταν κάτω από τις συνθήκε που σας περιέγραψα. Οπότε, από την άλλη μεριά το Target 2 είπατε ότι ανεβαίνει πάλι το εξηγήσαμε με τις πολιτικές μας ε, δράσεις, το οικονομικό μας δελτίο, ξανά και ξανά. Έχουμε εξηγήσει γιατί συνέβη πρόσφατα. Γιατί ως επιτοπλίστων συνδέεται με το πρόγραμμα αγορών. Το μεγαλύτερο μέρος του διακανονισμού των συναλλαγών αυτών, όπου μας πουλούν οι επενδυτές, τους τίτλους που αγοράζουμε. Ο διακανονισμός αυτός γίνεται από κοινού τις χώρες. Και έτσι κυκλοφορούν οι ροές και έτσι εξηγείται και η ισορροπία. Είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το συγκρίνουμε με την αύξηση του T2 κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπου υπήρξε πανικός, όπου υπήρξε κεφάλαια τα οποία έφευγαν από διάφορες χώρες. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στις αγορές. Οι τιμές, το ενεργητικό στις διάφορες χώρες έχουν προχωρήσει στη σταθεροποίηση τον τελευταίο καιρό. Άρα δεν πρόκειται για στρεσογόνα κατάσταση των αγορών. Έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι πληρωμές μας και κυρίως στη Γερμανία. Ευχαριστούμε. Άννα Μιράντα... όχι. Ο Σβέν Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κωνσταντσιο, ήθελα κι εγώ απλώς να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να σας πω αντίο, τουλάχιστον από θεσμική σκοπιά, διότι θυμάμαι καλά, όταν πρώτον αλάβατε τα καθήκοντά σας και όλη αυτή την οκταετία, το διάλογό μας και θέλω να σας θέσω ένα θεσμικού χαρακτήρα ερώτημα. Από τη μια τις τελευταίες εβδομάδες και μήνα είδαμε κάποιες, ε, κάποια σκάνδαλα ξεπλήματος βρώμικου χρήματο που μας φέρνουν σε δύσκολη θέση να ξεσπάνε στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα με μια τράπεζα που εποπτεύεται στην Λετωνία. Και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στη Λετωνία που δεν είναι ευχάριστο να τα ακούει κανεί να τα διαβάζει με την Φίνσεν και την Αμερικανική εμπλοκή. Οι Αμερικανικές αρχές κατά του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος άρχισαν να κάνουν εποπτεία στην Ευρώπη στην ουσία. Και απ' την άλλη, και με τη δική σας βοήθεια, δημιουργήσαμε τον ε, μηχανισμό αυτό για την παρακολούθηση της φοραπάτης και είδαμε κατά πόσον ε, πόσο πολύ μάλλον αναρωτιούνται οι άνθρωποι αν πρέπει να ανήκει στην ΕΚΤ και αν μπορεί να συνάδει με την εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Για την ώρα δεν έχει τη μεγαλύτερη ε, αξιοπιστία η εποπτική λοιπόν αρχή. Γιατί να μην γίνει η αρχή, η αλλαγή μάλλον, η μετατόπιση. Έχετε πολλές πληροφορίες για τρίτες χώρες με σημαντικές ροές χρήματος δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι παραπάνω για την εποπτεία σε περιπτώσει ξεπλημματο δρομικού χρήματο και με τι τόσο συνδέσεις που έχετε με τράπεζες και κυρίως να ελαφρύνεται τη δουλειά του, της εποπτικής αρχής για να ξεπεραστεί η ενδεχόμενη σύγκρουση αρμοδιοτήτων ή συμφερόντων με τον καθορισμό τη νομισματική πολιτική. Γιατί δεν γίνεται κάτι από θεσμική λοιπόν πλευρά. Ήδη βλέπω από την έκφρασή σα ότι δεν συμφωνείτε, αλλά πείτε μου πραγματικά τι πιστεύετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκίγκολτ. Να σας πω ότι και εγώ κατά τη διάρκεια των ετών έχω ε, ε, ε, βρει πολύ ικανοποιητικές τις ανταλλαγές απόψεων που είχαμε για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος. Όπως σας ε, υπόθηκε πρόσφατα στην ΕΚΟΝ από εκπροσωπό μας, δεν έχουμε αρμοδιότητα για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος, διότι υπάρχουν εθνικές αρχές υπεύθυνε γι' αυτό. Και έχουν μάλιστα και ανακριτικές αρμοδιότητες που εμείς δεν τις έχουμε. Έστω και αν είμαστε επόπτες. Άρα οι επόπτε και πολλοί κόσμοι δεν το καταλαβαίνει αυτό. Μπορούν να πάνε σε μια τράπεζα, να κοιτάξουν τα βιβλία του, αλλά αυτό που ελέγχουν είναι αυτό που του επιτρέπουν οι τράπεζε να ελέγξουν. Δεν έχουν αστυνομικό ένταλμα ή αρμοδιότητα να ε, ε, έχουν πρόσβαση στα αρχεία των υπολογιστών, να ελέγξουν άλλα αρχεία. Αυτά είναι ανακριτικέ αρμοδιότητε που δεν βρίσκονται στα χέρια των εποπτών. Οι επόπτε εξετάζουν και ελέγχουν ό,τι μπορούν. Ξέρετε όμως ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί κανείς να το ελέγξει μόνο από, με τις ε, συναλλαγές, της ροές χρήματος από μια τράπεζα σε μια άλλη. Το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος διαφαίνεται μόνο όταν η τράπεζα εφαρμόζει την αρχή του, της ταύτισης, της ταυτοπροσωπίας του πελάτη, δηλαδή να δει ακριβώς από πού προέρχεται ακριβώς το χρήμα. που μπορεί να έχει προκύψει από λαθρές ε, δραστηριότητε στη μαύρη αγορά. Όταν τότε το χρήμα ε, κατατεθεί σε μια τράπεζα, μπει ω κατάθεση σε μια τράπεζα, μπορεί μετά να φύγει για νόμιμες πληρωμές, νόμιμες συναλλαγές. Αυτό είναι το ξέπλυμα. Χρήμα που είναι εκτός του νομικού κυκλώματος, του επισήμως νομίμου μάλλον κυκλώματος, μπορεί μέσω κατάθεσης να φτάσει σε μια τράπεζα. Αυτό είναι το όλο Η αρχή της ε, ταυτοπροσωπείας ενός πελάτη, του να γνωρίζουν δηλαδή τον πελάτη, είναι ένα θέμα του κατά πόσο εφαρμόζεται. Αυτή είναι μια συμπεριφορά που μπορεί να ελεγχθεί και να εξεταστεί από τους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα να το κάνουν. Έτσι έχει κατάσταση με τα στατιστικά στοιχεία, με όλα τα δεδομένα με τις συναλλαγές από μια τράπεζα σε μια άλλη, που είναι και οι δύο δεν μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει τίποτα, απολύτως τίποτα για το ξέπλυμα. Γι' αυτό και παρεμπιπτόντως, οι Αμερικανικές αρχές που εντόπισαν την υπόθεση αυτήν το άλλων, δεν ε, κοίταζαν τις ροές χρημάτων, χρήματος, άλλου τρόπο βρήκανε και είναι και αυτό κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου. Πιστεύουμε πάντως, εγώ συγκεκριμένα δηλαδή, το ευρωπαϊκό σύστημα με τις εθνικές αρχές να είναι αρμόδιες για τα θέματα αυτά του ξεπλήματος δεν είναι καλό. Θα έπρεπε να υπάρξει μια κεντρική διοργάνωση ή επιβολή υποχρεωτική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο επίπεδο του δικτύου αυτών των εθνικών αρχών για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Θα έπρεπε κάποια στιγμή να ληφθεί αυτή η απόφαση, γιατί είναι σημαντικό να βελτιώσουμε τι δυνατότητε διερεύνηση. Τώρα για την ε, υποπτική αρχή, την αρχή υποπτήση των τραπεζών. Δημιουργήθηκε η αρχή αυτή, αλλά έχουν συμβεί τα εξή δύο από τη στιγμή τη ίδρυσή τη. Πρώτα απ' όλα το Brexit Όπως τα γνωρίζετε, μόλις ε, αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, τα συνολικά, τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 97-98% θα εμπίπτουν στο μηχανισμό ε, σταθερότητας που είναι μέρος των αρμοδιοτήτων της ΕΚΤ και της Τραπεζικής Αρχής. Η ΕΚΤ ανέλαβε λοιπόν αυτέ τις αρμοδιότητες που δεν είχε στην αρχή και μετά το Brexit το 97-97% των ενεργητικών ε, στοιχείων των τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ε, στα δικά μα χέρια. Και η απόδοση αυτών των αρμοδιοτήτων στην ΕΚΤ σημαίνει ότι ουσιαστικά γίναμε και αρχή προς τις μακροπροληπτικές πολιτικές και αρχές. Άρα πρόκειται για μια κατάσταση που διαφέρει. Και γι' αυτό, λόγου χάρη, ε, σε αντίθεση με τη δική σας την άποψη, μια από τις ε, πρώτες εφημερίδες είπε ότι το καλύτερο ήταν να ε, ενταχθεί η εποπτική αρχή στην ΕΚΤ για να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις νέες συνθήκες. Ακριβώς το αντίθετο συμπέρασμα αυτό στο οποίο καταλήγετε εσείς. Η Εποπτική Αρχή για τις Τράπεζες μόνο προειδοποιήσεις μπορεί να εκδώσει. Δεν μπορεί να επιβάλλει τίποτα σε κανέναν με μια τελεσίδικη απόφαση. Μόνο προειδοποιήσεις και συστάσεις. Και ίσως γι' αυτό να θεωρείτε ότι δεν ήταν πολύ αποτελεσματική στη δράση της, αλλά προειδοποίησεις έχει εκδώσει. Κάποιες φορές δεν ε, ακολουθούνται από δράση, δεν έχουν κάποιο αντίκτυπο χειροπιαστό, αλλά αυτή είναι η δουλειά της. Τώρα, αυτές οι εξελίξεις πρέπει να εξεταστούν από την εξή σκοπιά. Θα πρέπει να, να γίνει κατανοητό ότι η μακροπροληπτική μα αρμοδιότητα, όπως έχει προκύψει μέσα από την οπτική αρχή των είναι κάτι που πάντα το και η νομοθεσία, που δεν έχει γίνει ακόμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο Γκουαλτιέρη. Για την SRP βέβαια είμαι κάπως επιφυλακτικός. Έχουμε ήδη αρκετούς θεσμούς, αρκετά θεσμικά όργανα. Προσθέσουμε κι άλλο ένα ίσως οδηγήσει σε μεγαλύτερη σύγχυση. Αυτή είναι η ε, γνώμη μου. Μαρίζα Ματίας τώρα ακολουθεί, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την τελευταία ανταλλαγή απόψεων που έχουμε στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Όλα αυτά τα χρόνια μας βοηθήσατε στην Επιτροπή μας και ήσασταν πάντα διαθέσιμος για να συζητάμε τις διάφορες προοπτικές. Ήθελα να θέσω ένα θέμα που κι άλλες φορές το έχω θέσει στα πλαίσια αυτού του διαλόγου και την τελευταία φορά, αλλά θα ήθελα να εμβαθύνουμε λίγο. Είναι ο ρόλος της ΕΚΤ στην αγορά και ομολόγων από τις διάφορες χώρες. Όχι που βρίσκονται υπό κάποιο πρόγραμμα εξυγίανσης ε, που μπορεί να το έχουν ολοκληρώσει. Η πώληση ομολόγων από την ΕΚΤ έχει δυσκολέψει τις μακροοικονομικές τους προοπτικές θα, δω, θα δούμε βεβαίω εάν μπορούμε να έχουμε πραγματικέ απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα. πάντω, η ΕΚΤ ουσιαστικά μετέφερε τα χρέη των περιφερειακών χωρών προς το κέντρο. Το ερώτημα λοιπόν είναι αν θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε, να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό που εδώ και χρόνια έχουμε δει να ανακύπτει, θα το δεχθούμε ως ένα απετελεσμένο γεγονός ή η ΕΚΤ ουσιαστικά εμέσως πριν σαφώς ε, επιτρέπει τη μεταφορά κεφαλαίων από την περιφέρεια προς το κέντρο εντείνοντας έτσι τις ε, υπάρχουσες μακροοικονομικές ανισότητες και έπειτα για το νέα προεδρία της ΕΚΤ και τις νέες ε, αντιπροεδρίες, δηλαδή όσους θα αναλάβουν νέα καθήκοντα στην ΕΚ, της επίπεδο Προέδρου και Αντιπροέδρου. Ήθελα να μου πείτε αν αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια αγγίηση ότι μπορεί να υπάρξει μια μακροπόθεσμη συμφωνία για την νομισματική πολιτική της ΕΚΤ ή αν μπορούμε να περιμένουμε εκπλήξεις Θα απαντήσω αγγλικά για διευκόλυνση των υπολείπων. Για την πρώτη σας ερώτηση δεν συμφωνώ, όπως καταλάβατε και από τις κινήσεις μου και τις εκφράσεις μου. Με συγχωρείτε κιόλα. Αλλά λέτε ότι αυτό ήταν τρομερά επιζήμιο για τις χώρες αυτές. Σχεδόν, δεν το είπατε έτσι, αλλά σχεδόν Καλύτερα θα ήταν να μην έχουμε καν ανάμειξη. Ναι, ναι, δεν το εννοήσατε, δεν το είπατε, αλλά ήσασταν κάπως κατηγορηματικοί ε, στο να κατηγορείτε τη μεταφορά κεφαλαίων ως αποτέλεσμα των προγραμμάτων που επιβλήθηκαν ε, στις χώρες. Ε, το ερώτημα δεν είναι ακριβώς όπως το θέσατε εσείς. Η ΕΚΤ είναι απλώς μία συνιστόσα του ευρωσυστήματος. Τα ποσοστά Οι μεταφορές δεν έγιναν από την ΕΚΤ. Οι, αγορές, οι εξαγορές χρέους δεν έγιναν από την ΕΚΤ, έγιναν από άλλα ιδρύματα και τα κέρδη, τα έσοδα από αυτές τις ε, συναλλαγές έμειναν στα χέρια των εθνικών κεντρικών τραπεζών, στους δικούς τους λογαριασμούς, στα δικά τους βιβλία και τα διένυμαν στους ε, πελάτες τους, τους μετόχους τους, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία. Η ΕΚΤ επίσης αγόρασε ένα μικρό μέρος αυτών ε, αξιογράφων. Και ως προς τα κέρδη, ως προς το κεφάλαιο και να ανοίξω μια παρένθεση λέγοντας ότι σε αντίθεση με πολλές απόψεις που ακούστηκαν τότε, η ΕΚΤ δεν, δεν μετατράπηκε σε μια κακή τράπεζα με τοξικά ε, περιουσιακά. Δεν ισχύει γιατί δεν ήταν καθόλου τοξικά, υπήρξαν κέρδη όπως είπατε. Αυτό Έγινε όμως σε όλα τα παρακλάδια του ευρωσυστήματος, άρα και στην ΕΚΤ. Τώρα, τι γίνεται με τα έσοδα που έχει η ΕΚΤ, με τα κέρδη. Μπορούμε να ενισχύσουμε το κεντρικό μας αποθεματικό, αλλά μόνο μέχρι εκεί που επιτρέπει το κεφάλαιο της ΕΚΤ. Δεν μπορούμε δηλαδή να το ενισχύσουμε χωρίς όριο, ήδη έχουμε φτάσει στο ανώτατο. Το, το, κέρδο, το κέρδος που περισσεύει ξαναδιανέμεται στις κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών, στις εθνικές κεντρικές τράπεζες που με τη σειρά τους τα δίνουν στις κυβερνήσεις τους. Δεν υπήρξε λοιπόν κάποια τεράστια μεταφορά από την περιφέρεια και άλλες χώρες προς το κέντρο, την ΕΚΤ. Σας το εξήγησα με αυτήν την ε, ανάλυση και μετά το κέρδος από όλα αυτά ξαναποδόθηκε στις κυβερνήσεις. Όχι βεβαίως ε, ένα προς ένα, αλλά αναλόγως με τον συνολικό υπολογισμό. Την, ε, την κατανομή του κέρδους την φροντίζουν μετά οι εθνικές κεντρικές τράπεζες. Αλλά όλες οι κεντρικές τράπεζες του ευρωσυστήματος είχαν κέρδος και έδωσαν τα μερίσματα στους μετόχους τους. Και αυτό ως αποτέλεσμα του κέρδους από τα σχετικά προγράμματα. Επίσης σκεφτείτε ότι και οι και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες πρέπει να είναι χρηματοοικονομικώς ε, εύρωστες στους ισολογισμούς τους. Αυτό και ως αποτέλεσμα των όσων ορίζει η συνθήκη. Αλλά το θέμα είναι τι μπορεί ο κέρδο να ενταχθεί στο γενικό μα αποθεματικό και τι πρέπει να αποδοθεί πίσω στις εθνικέ κεντρικέ τράπεζε. Για το δεύτερο σα ερώτημα, Νομίζω ότι μπορεί και να έχετε περισσότερο ε, επιρροή στο τι θα γίνει στο μέλλον με τις θέσεις του Πρόεδρου και του Πρόεδρου στην ΕΚΤ, από εμείς οι ίδιοι στην ΕΚΤ. Έχετε ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε εδώ στις μελλοντικέ επιλογές. Thank you, James Ευχαριστούμε, κύριο Κόμπερν. όχι ακριβώ James Coburn, αυτό ήταν ένα σπουδαίο ηθοποιό που είχε παίξει και στου 7, ήταν υπέροχη. Χαίρομαι πάντω που σα βλέπω, λέγομαι David. Χαίρομαι που σας ε, βλέπω. Η Deutsche Bank και η περίπτωσή τη είναι εξαιρετικά ανισχυτικά. Είμαι βέβαιο ότι και εσείς ανισχύετε το ίδιο όπω και εγώ. Οι Ιταλικέ τράπεζε εξάλλου και αυτέ φαίνεται να μην τα πηγαίνουν καθόλου καλά, μάλλον τρομακτική είναι η κατάστασή του. Έχω ξαναρωτήσει και άλλες φορές άλλους την ερώτηση αυτή. Δεν νομίζετε ότι οι κύριοι Βερχόφστατ και Μπαρνιέ που προσπαθούν να επιβάλλουν κυρώσεις, να τιμωρήσουν δηλαδή το ΣΥΡΙ του Λονδίνου ότι δεν είναι απόλυτα σόφρον η στάση τους αυτή όταν τράπεζες και γερμανικές και ιταλικές ε, δεν φαίνεται τα πιούν καθόλου καλά. μήπως κάποια στιγμή ε, ανατραπούν οι ε, τράπεζες αυτές, δηλαδή ε, καταρρεύσουν οι τράπεζες αυτές επειδή δεν θα έχουν αρκετές πιστώσεις, επειδή δεν θα λειτουργεί το ΣΥΤ του Λονδίνου. Και τα πράγματα δεν θα πάνε καλά τότε. Μήπως θα πρέπει να μιλήσετε με αυτούς τους κυρίους Μπαρνιέ και Βερχόφστατ που πάνε λίγο να γίνουν ο χονδός και ο λιγνός του Brexit και να δείξουν κάποια μεγαλύτερη ευαισθησία για το μέλλον, ότι θα χρειαστεί δηλαδή να κάνουν business με το Λονδίνο και στο μέλλον. Ιδίω με ένα επιτυχημένο εταίρο όπως θα είμαστε εμείς, όταν οι τράπεζες οι δικές σας θα είναι τα χάλια τους. Ο κ. Κωνστάνσιο, ευχαριστώ. Δεν συμφωνώ με την πολύ αρνητική εικόνα που δίνεται των τραπεζών που αναφέρατε Έχω δίκιο, λέει ο κ. Κομπέλη. Καλά, θα το δούμε, απαντάει ο κ. Κωνστάσιο. Να σα πω όμω το εξή. Η ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών γενικά έχει βελτιωθεί σημαντικά, κατά μέσον όρο. Κατά μέσον όρο λοιπόν, ο λόγος μεταξύ δύο κεφαλαίου και μετοχών Common Equity είναι, άμα βάλετε και τα άλλα μέσα, φτάνει στο 18% και στο 19%. Ο αριθμός αυτός για την Common Equity Ratio ήταν στο 7% το 2007 και το έχει φτάσει στο 14,3%. 14,3. Υπάρχει λοιπόν πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα συνολικά. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο όμως ε, για το θέμα αυτό. Δεν συμφωνώ λοιπόν με την πολύ αυτή αρνητική εικόνα που δώσατε. Πράγματι, ορισμένε τράπεζε είναι σε πρόγραμμα, ε, έχουν προβλήματα. Και εσεί όμω στο Ηνωμένο Βασίλειο έχετε κάποια προβλήματα στι τράπεζε σα και αυτό ισχύει. Τώρα, να λέει όμω κανεί ότι η Ευρώπη τιμωρεί το ΣΥΤ του Λονδίνου. Δεν έχουμε εμεί απολύτω καμία σχέση με τη δική σα θεμητή άλλωστε απόφαση να αποχωρήσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποχωρήσετε και από την ενιαία αγορά. Ε, αυτά θα είναι οι συνέπειε των αποφασιών σα. Τι αποφάσει αυτέ τι έλαβε το Ηνωμένο Σύριο, δεν τι αναλάβε, δεν τι Ναι, ναι, αφήστε με να τελειώσω. Είμαι απολύτω βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε business με το Ηνωμένο Βασίλειο και σε σημαντικό βαθμό. Βιομηχανικά αγαθά θα πηγαίνουν έρχονται, χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε και ούτω καθεξή. Ναι, βεβαίω. Αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά αυτό το οποίο υπονοείτε δεν είναι αυτό. Εσείς υπονοείτε ότι παρόλο που θα είστε απέξως, παρόλο που θα έχετε τις δικές σας ρυθμίσεις, τη δική σας εποπτεία, τη δική σας παρακολούθηση των πιστοτικών συντριβάτων, εσείς ή θα να είσαστε λοιπόν απ' έξω, ταυτόχρονα να είσαστε όμως μέσα στην ενιαία αγορά τραπεζικών υπηρεσιών, σαν να μην βγήκατε ποτέ. Αυτό δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να μείνει κανείς. Ουδής επιθυμεί να τιμωρήσει το ΣΥΤ του Λονδίνου. Θα γίνουν συμφωνίες για να συνεχιστούν οι business, αλλά με κάπως διαφορετική βάση. Αυτό είναι και το αναμενόμενο ε, φυσιολογικό αποτέλεσμα της ε, θεμητής σας απόφασης να αποχωρήσετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ έτσι το βλέπω το πράγμα. Δημοκρατική απόψη. Ναι, ναι. Που είναι το δικαίωμα του καθενός. Ναι. Ωραία. Τότε γιατί είστε τόσο αρνητικοί, επιμένει ο κ. Κομπέρν. Αφού αυτή είναι η απόφαση του Βρετανικού λαού, γιατί Εγώ δεν έδωσα στα λόγια μου απολύτως κανένα αρνητικό χαρακτήρα. Τι να πω, αυτά πέστε το βρετανικό κοινό. Γουαλτιέρη. Εσείς θέλατε να φύγετε από την... Αλλά μου φαίνεται τώρα σαν να θέλετε να μείνετε. Όχι, όχι, δεν θέλω, δεν θέλω. Speak Dutch. Um, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άνεμαντς. Επανέρχομαι στην ερώτηση Κλίντσεντ για το T2. Φαίνεται από τη δικιά σας την τοποθέτηση τουλάχιστον, μιλάτε για ένα κλειστό σύστημα. Ωραία, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα αλλά η ερώτηση που αφορά και πολλούς Γερμανούς συναδέλφους έχει να κάνει με αυτά που δημοσιεύθηκαν. μελέτη δηλαδή του Ινστιτούτου Φέρι, με έρευνα η οποία λέει ότι με τίποτα δεν πρόκειται να υπάρξει κατάρρευση. Υπάρχει το σχέδιο του κύριου Μακρόν για μεγαλύτερη ένταξη και υπάρχει και ακριβώς το Target 2. Στο σύστημα αυτό λοιπόν που θέλουμε να επανέλθει σε μια κανονική κατάσταση είναι ένα σύστημα το οποίο όμως καταχραστήκαμε για πολύ καιρό όσον αφορά χώρες δηλαδή η Γερμανία, Λουξεμβούργο σε μικρότερο βαθμό η Ολλανδία, ε, η Ισπανία, η Ελλάδα σε λιγότερο βαθμό η Πορτογαλία με πολλά δισεκατομμύρια. Ρωτώ λοιπόν, αν υπάρξουν προβλήματα, αν δηλαδή χρειαστεί να βγει από την Ευρωζώνη μια χώρα, τι θα γίνει αν ισχύουν αυτά τα οποία προβλέπει και το Ινστιτούτο φέρει. Όπως είπα και στην προηγούμενη απάντησή μου, ό,τι προβλήματα μπορεί να έχουν ε, με αυτούς τους λογισμους ότι δύο, μπορεί να προκύψουν εφόσον μία χώρα είναι να βγει από την Ευρωζώνη. Και νομίζω ότι είναι αρκετά πίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι. Θα ήταν ε, πρώτα απ' όλα ιδιαίτερα δραματικό για την ίδια τη χώρα, όποια χώρα και αν είναι αυτή. Και σύμφωνα με τις ηθίκες, καμία χώρα δεν μπορεί να εκδιωχθεί έτσι. Πρέπει δηλαδή να την πάρει την απόφαση η ίδια η χώρα ότι θέλει να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο. Στη συνέχεια, αναφέρεστε σε δάνεια. Εδώ όμως δεν πρόκειται για δάνεια. Στις χώρες αυτές, οι οικονομικοί παράγοντες των χωρών αυτών δημιούργησαν ευρώ χωρίς χρήματα από την ε, Κεντρική Τράπεζα. Δεν δίνει επιστώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έτσι στον κόσμο. Οι οικονομικοί παράγοντες δημιούργησαν τα ευρώ, αλλά έπρεπε βέβαια να τα πληρώσουν τα ευρώ σε κάποιον άλλον, σε κάποια άλλη χώρα. δεν πήραν δάνεια από την Κεντρική Τράπεζα για να αποκτήσουν αυτά τα ευρώ. Υπήρξαν τα νοικοκυριά, υπήρξαν επιχειρήσεις, οπότε τα ευρώ αυτό πάνε στην άλλη χώρα μέσα από το σύστημα των κεντρικών τραπεζών. Αυτή είναι η κανονική κυκλοφορία, άπαξ και έχεις ένα κοινό νόμισμα. Οπότε είναι αναπόφευκτο ότι αυτό οδηγεί στην κυκλοφορία του νομίσματος που χρησιμοποιούν τώρα οικονομικοί παράγοντες σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Η οργάνωση δηλαδή αυτής της διαδικασίας είναι τέτοια που προβλέπεται η καταγραφή αυτών ε, των ε, ισολογισμών ε, στις τράπεζες των διαφόρων χωρών μελών. Και είπαμε, αν μια χώρα ήταν να βγει από την Ευρωζώνη, τότε θα υπήρχαν πιστώσεις, αλλά όπως είπα και πριν, η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει το ενεργητικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ευθύνε της. Είναι μια αναπόφευκτη συνέπεια δεδομένου ότι έχουμε μια νομισματική ένωση, έχουμε ένα ενιαίο νόμισμα. Έτσι είναι. Αλλά όπως επίσης είπα, αυτή τη φορά η αύξηση του target του balances δεν έχει να κάνει με μια στρεσογόνα κατάσταση, με διαφυγή κεφαλαίων ε, από χώρες κτλ. Το έχουμε δείξει στις ε, δημοσιεύσεις μας ποια είναι η τάση και ποιος είναι ο διακανονισμός για τις συναλλαγές που κάνουμε, αγορές κτλ. Αυτό μπορώ να σας πω για το target του και το πώς λειτουργεί. Ευχαριστούμε. Γαβριέλ Μάτο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε Κωνσταντιο Χαίρομαι που είσαστε εδώ μαζί μας σήμερα. Ξέρετε και το είπατε ότι στηρίζουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και την νομισματική πολιτική, ξέροντας βέβαια ότι δεν φτάνει για μια σταθερή ανάκαμψη. Επανέρχομαι στον πληθωρισμό. Είπαμε ότι αυξήθηκε, κάτω είναι πάντα από τον στόχο μας, όπως το εξηγήσατε και εσείς πολύ καλά. Και βλέπουμε ποιες είναι οι προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και η ΕΚΤΑ συζητώντας το θέμα της προσωπικής χαλάρωσης, κατά πόσο θα επεκταθεί ή όχι. Εσείς μας λέτε ότι σιγά σιγά θα σταματήσει. Λοιπόν, θέλω να ξέρω τι χρονοδιάγραμμα προβλέπει η τραπεζά σας και τι θα γίνει με τις χώρες της Ευρωζώνης. Και κάτι άλλο που μερικές φορές δεν μας καταλαβαίνουν οι πολίτες. Εγώ θα ήθελα να τα λέμε πιο ξεκάθαρα για να μας καταλαβαίνουν. Η αύξηση της ανάπτυξης και η νομισματική πολιτική δεν ερμηνεύονται σε σταθερή αύξηση και του πληθωρισμού. Οπότε, για ποιους λόγους και ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση, ώστε να μην μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας για τον πληθωρισμό με τρόπο που να καταλαβαίνουν οι πολίτες. Γιατί οι πολίτες πέρασαν από την κρίση, πέφεραν από αυτήν και θα ήθελαν να μπορούν να καταλάβουν. Λέμε ότι ξεπεράστηκε η κρίση και μιλάμε για ανάκαμψη. Όμως ο κόσμος αυτό δεν το νιώθει. Ένιωσε την κρίση, αλλά δεν αντιλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο όπως αντιλήφθηκε την κρίση το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ανάκαμψη. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε τι μήνυμα μπορούμε να στείλουμε στο κόσμο που ζει δύσκολα αυτές τις εποχές για να καταλάβετε ότι βρισκόμαστε σε ανάκαμψη και ότι η κρίση αρχίζει να είναι παρελθόν. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Θα αρχίσω με το πρώτο στοιχείο της ερώτησής σας. Εγώ δεν βλέπω η σταδιακή προσαρμογή του προγράμματός μας ε, αγοράς μη συμβατικών μέτρων να μπορεί να είναι κάτι αρνητικό για την ανάπτυξη. Όχι. Κάνουμε προσαρμογές και γιατί, ακριβώς γιατί υπάρχει ανάκαμψη, όπως είπατε ότι είναι πραγματικότητα. Πέρυσι είχαμε 2,5% ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Στις προβλέψεις μας έχουμε 2,4% για φέτος και 2,9% για του χρόνου. Οπότε υπάρχει ανάκαμψη. Παρόλο που η ανεργία είναι ψηλή, ο μέσος όρος είναι 8,5 που είναι το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008 και μετά. Άρα υλοποιείται η ανάκαμψη. Και δεν λέω ότι σε όλους τους τομείς της κοινωνίας ή ότι όλοι οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται την ανάκαμψη αυτή. Αν δείτε τις ε, εξελίξεις, τους δείκτες, αν ε, δείτε, κατά μέσο όρο βέβαια πάντα, έτσι, ε, την κατανάλωση των καταναλωτών, την αισιοδοξία των καταναλωτών, διαπιστώνετε ότι υπάρχει κάτι θετικό. Υπάρχει αυτή η ανάκαμψη, δηλαδή γίνεται αισθητή στους καταναλωτές γενικά. Η ιδιωτική κατανάλωση ήταν και ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην ανάκαμψή μας. Από πλευράς δαπανών δηλαδή που αυξήθηκαν η ιδιωτική κατανάλωση. Αυτό δείχνει ότι πολλοί καταναλωτές είχαν χρήματα στα χέρια τους και αύξησαν τις αγορές τους. Όλα αυτά αποτελούν δείγματα. Βέβαια, συμφωνώ μαζί σα ότι σε πολλέ κατηγορίε του πληθυσμού και σε κάποιε χώρε περισσότερο από ό,τι σε άλλε, ε, κάποιοι δεν έχουν αντιληφθεί καμία ανάκαμψη. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά είναι η ίδια η φύση της κατάστασης και ο τρόπος που λειτουργούν οι οικονομίες μας, που είναι οργανωμένες οι οικονομίες μας στις διάφορες χώρες. Αλλά δεν είναι σωστό να λέτε ότι οι καταναλωτές δεν έχουν νιώσει την ανάκαμψη καθόλου. Οι μισθοί, εντάξει, είναι πολύ περιορισμένοι ακόμα, πράγματι, και αυτό μας εκπλήσει, γιατί εμείς περιμέναμε ότι με την ε, ανάπτυξη, την οικονομική, θα υπήρξε και αύξηση των μισθών. Κάποια τέτοια δείγματα υπάρχουν αλλά προς το παρόν δεν είναι πολύ πιστικά. Και σίγουρα είναι χαμηλότερα από τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε για την Ευρωζώνη. Και πάλι λέω, είναι περίεργο, γιατί ενώ έχουμε ανάπτυξη δεν αυξάνονται μισθοί. Πολλέ είναι οι εξηγήσει. Πρώτα απ' όλα η αδράνεια από την κρίση, που έχει σαν αποτέλεσμα να είναι όλοι πολύ πιο προσεκτικοί στο πώ συμπεριφέρονται και έτσι πράγματι τα σεδικάτα, οι εργαζόμενοι ε, φαίνεται να δέχονται. Γιατί φοβούνται μην χάσουν τη δουλειά τους, έτσι μην ε, έχουν ε, περισσότερη ενέργεια, Δέχονται λοιπόν να μην αυξάνονται τόσο πολύ οι μισθοί τους. Οπότε αυτή η αδράνεια είναι μια εξήγηση. Θα αλλάξει, έτσι είναι θέμα χρόνου για να αλλάξει. Επίσης υπήρξε και το θέμα του νομίσματος, η άνοδος. Όλα αυτά εξηγούν τις εξελίξεις. Πάντως τα νούμερα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Συνεπώς, ελπίζουμε με ανακατανεμικές πολιτικές θα τα καταφέρουμε. Και αν συνεχίσει η αύξηση της απασχόλησης, θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες και για τους τομείς εκείνους της κοινωνίας που δεν έχουν ακόμα ε, αντιληφθεί επαρκώς την ανάκαμψη. Δεν την έχουν νιώσει οι ίδιοι. Πάντως από το 2014 είμαστε η μόνη περιοχή του κόσμου που δημιούργησε πάνω από 6 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Ε, αυτό κάποιος το νιώθει. Και σας είπα ότι οι καταναλωτές ε, γενικά καταναλώνουν περισσότερα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη, οπότε είναι και αυτό ένα δείγμα. Ευχαριστούμε κύριος Περέιρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να ξεκινήσω χαιρετίζοντα ε, τον ε, κύριο Κωνστάντσιο για αυτή την τελευταία παρουσία εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο επειδή ήταν ένας αξιόλογος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ και συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας που έδωσε αξία και νόημα και στο θεσμό με τη δουλειά του. Τον ευχαριστούμε και για την ε, συνεργασία και την κοινωνία που είχε με το Ευρωκοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της οκταετούς του θητεία Το 2017, όπως υπενθυμίστηκε εδώ, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και αφού αποφύγαμε την κατάρρευση της Ευρωζώνης, όπως υπόθηκε προηγουμένως, καταφέρατε εσείς να διατηρήσετε έναν καθοριστικό ρόλο στην σταθεροποίηση της Ευρωζώνης και την συνεργασία των οικονομιών. Και σε αντίθεση με τα επικριτικά σχόλια που έγιναν εδώ από τον γερμανό συνάδελφο του ΕΛΚ, του κυρίου Μπούλτς, Μπάλτς μάλλον, συγγνώμη, ε, εδώ είδαμε σύνεση στην νομισματική πολιτική της ΕΚΤ και την ε, ε, εξέλιξή της με την διάθεση της εξομάλυνσης και την ανάληψη ευθύνης. Διότι ο στόχος του πληθωρισμού που είναι ένα κεντρική σημασία πεδίο της ΕΚΤ είναι κάτι που πρέπει να επιτευχθεί και έχει επιτευχθεί εν μέρη ε, με τρόπο βιώσιμο για έναν τουλάχιστον προβλέψιμο ορίζοντα. Ήθελα να κάνω πάντως δύο ερωτήσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με τη μακροοικονομική πολιτική. Ακόμα και διατηρώντας μια νομισματική πολιτική, τουλάχιστον για λίγο καιρό ακόμα, ε, προς την υποστήριξη της οικονομίας, είναι φυσικό να μην διαρκέσει για πάντα. Αυτό που με απασχολεί είναι κατά πόσον βλέπετε να υπάρχει τάση μιας σταδιακής ανάκτησης της νομισματικής πολιτικής και αν αυτό είναι ένας επιπλέον παράγοντας να απαιτήσουμε τη συμβολή και άλλων πολιτικών, κυρίως των διαστατικών πολιτικών και πάνω απ' όλα των δημοσιονομικών πολιτικών. Και όλος ιδιαίτερος, εάν σημαίνει αυτό ότι η δημοσιονομική πολιτική που ήταν ουδέτερη τα τελευταία χρόνια ε, θα πρέπει να μετακινηθεί με κάθε υπευθυνότητα βεβαίως αλλά με μεγαλύτερη συμβολή των χωρών που έχουν περισσότερο δημοσιονομικό περιθώριο. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τις μεταρρυθμίσεις της Ευρωζώνης. Εδώ μας ε, φέρατε ένα μήνυμα υπέρ της Τραπεζικής Ένωσης. Αυτό που ήθελα να σημειωθεί είναι ότι αν υπάρχει ένας κατάλογος προτεραιοτήτων για την μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης και αν ε, λαμβάνεται υπόψη η δημοσιονομική δυνατότητα των χωρών. γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό θα έχουμε πάντα μια εξελαχίστων ε, κατάρτιση προτεραιοτήτων χωρίς να προχωρούμε. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω στα αγγλικά για να καταλάβουν ε, περισσότεροι στο κοινό. Ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια. Και όσο είπατε για την ε, δουλειά μου. Για τις ερωτήσεις σας. Η νομισματική πολιτική έχει να κάνει και με την καλή εξέλιξη της οικονομίας και θέλουμε εξομάλυνση, αλλά δεν είναι ο στόχος να γίνουμε πιο περιοριστικοί αν γίνουμε αν, γίνουμε πιο αν γίνουμε πιο περιοριστικοί, θα έχει να κάνει με το πώ εξελίσσεται η κατάσταση. Τα χρόνια που πάνε καλά τα πράγματα, τα επιτόκια αυξάνονται και αυτό μπορεί να αυξάνει την αγοραστική δύναμη κάποιων. Εάν αυξηθεί κι άλλο, μπορεί να, αυξηθεί και, να αυξηθούν και οι δυνατότητέ μα. Στο ε, ΑΕΠ, σε στους αριθμούς τουλάχιστον του ΑΕΠ, ε, Πάντως, για τη δημοσιονομική πολιτική μπορεί κανείς να πει όντως ότι η δημοσιονομική πολιτική χρειάστηκε να προσαρμοστεί στην κατάσταση και να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. δεν υπάρχουν κραδασμοί τρίχνοι που μπορεί να προκύψουν ξαφνικά, η όλη η δημοσιονομική πολιτική θα ε, χρειαστεί να προσαρμοστεί ε, απαραίτητο, ε, αναλόγως, όπως έγινε και στην περίοδο της κρίσης. Και όντως η ερμηνεία της Επιτροπής του 2015 και 2016 για την ευελιξία του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη σε περιπτώσει όπου υπάρξουν τριγμοί ή δυσκολίε, είναι κάτι που πλέον το επιτρέπει. Καθώ και η χρήση του δημοσιονομικού περιθωρίου που έχουν τα διάφορα κράτη-μέλη. Όμως μπορεί κανείς να πει ότι εάν στο μέλλον, όχι το απότερο μέλλον, δεν είναι κάτι το εντελώς απίθανο, ε, αλλά αν υπάρξει κάποιο νέο σοκ, κάποια νέα έφυση, θα πρέπει να ε, υπολογίσουμε περισσότερο στην δημοσιονομική πολιτική και να ελπίζουμε ότι θα αντιδράσει σε τέτοιο τριγμό, τέτοιο κραδασμό. Για τη δεύτερη ε, ερώτησή σας, ευκαιρία να απαντήσω συμπληρωματικά και σε έναν από τους συναδέλφους σας, για αυτά που πρότεινε ο πρόεδρος Μακρόν. Ναι, εσείς είσαστε. Αλλά πριν ε, κάνει αυτές τις προτάσεις ο πρόεδρος Μακρόν, η δημοσιονομική δυνατότητα ήταν κάτι που το ανέφερε και η έκθεση των πέντε πρόεδρων. Ήδη από το 2015. Και αυτό για μένα ήταν σημαντική συνιστόσα ε, για να συνυπολογιστεί στι μελλοντικέ μεταρρυθμίσει τη Ευρωζώνη. Για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ασυμμετρικού κατασμού και συμμετρικού. Πρόκειται για μια λειτουργία μακροοικονομική σταθεροποίηση που απαιτείται για την Νομισματική Ένωση. Και αυτό, κατά την άποψή μου, και εδώ μιλώ τελείω προσωπικά, κατά την άποψή μου δεν είναι θέμα της ε, ακριβώς αντίστοιχης και ίσης χρήσης δημοσιονομικών γραμμών για την Ευρωζώνη είναι η χρήση κονδυλίων όταν θα υπάρξουν σημαντικοί μακροοικονομικοί κραδασμοί για να συμβάλλουμε στη θεσταροποίηση της ε, μακροοικονομικής κατάστασης. Ναι, και για την νομισματική ένωση, κάτι που δεν πετύχαμε και πρέπει να το ε, επιζητήσουμε, είναι η ανθεκτικότητα. Είναι σημαντικό η ανθεκτικότητα αυτή να επιτρέψει να λειτουργήσει πιο ομαλά και χωρίς διακοπές η Νομισματική Ένωση. Αλλά αυτό θα γινόταν εάν αποφεύγαμε τον κατακαιρματισμό. Όπως Γκουαλτιέ, ευχαριστώ. Τώρα για τους τελευταίους ομιλητές θα παρακαλέσω να σεβαστούν όλοι το χρονικό όριο. Γαβριέλ Μάτο. Ναι, να αλλάξω λίγο θέμα. Κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει είναι στη λήξη της θητείας μας να προχωρήσει η Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και γι' αυτό και μιλάμε και για ίδια δημοσιονομική ικανότητα. Υπήρξε δημοσίευση πρότασης για να σχεδιαστεί ένας κεντρικό μηχανισμός σταθεροποίηση που να αντιμετωπίσει τα σύμμετρα σοκ στι διάφορε χώρε μέλη. Και η πρόταση, αν κατάλαβα καλά, έχει ιδιαίτερη σημασία για κάποιου οικονομικούς για οικονομικούς τομεί μιλάει και όχι για χώρε συγκεκριμένα. Γιατί στόχο ε, της ΕΚΤ είναι ακριβώ να μην δημιουργήσει έναν μηχανισμό αυτόματης μεταφοράς από μία χώρα στην άλλη. Η ερώτηση λοιπόν είναι πώς θα διασφαλίσουμε αυτό το επίπεδο για να λειτουργήσει καλά επικεντρωμένη σε συγκεκριμένους οικονομικούς ε, τομείς, αλλά και σε χώρες αν βρεθούν σε ανάγκη πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο μηχανισμό σταθερότητας που να διασφαλίζει σε αυτές τις χώρες της Ευρωζώνης όταν βρίσκονται σε κρίση ότι θα μπορέσουν να βοηθηθούν. Πρώτον, η ΕΚΤ ως θεσμικό όργανο δεν έχει δημοσιεύσει καμία συγκεκριμένη πρόταση για το πώς θα είχε αυτό το κεντρικό όργανο. Έχουμε τις προτάσεις ε, των αντιπροέδρων, ε, πώς θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο, αλλά τις λεπτομέρειες δεν τις έχουμε. Δεν έχουμε δεσμευτεί προς καμία συγκεκριμένη πρόταση. Θα υπάρξει ένα ε, σχέδιο, ένα έγγραφο εργασίας, το οποίο όμως δεν δεσμεύει θεσμικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Πολλές λύσεις υπάρχουν για αυτήν την ε, μακροπρόθεσμη σταθερότητα ε, με πληρωμές από το κέντρο, με άλλες χρηματοδοτήσεις, από κάποια γραμμή, από προστασία των επενδύσεων. Πολλές λύσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ενδεχομένω, αλλά δεν υπάρχει τίποτα επίσημο θεσμικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπέρ της μακροσταθερότητας. Ο κύριος Φων Βάιτσεκερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, μεγάλη χαρά που σας βλέπω πάλι. Πρώτη ερώτηση. Σας ερωτώ για πράγματα που έγιναν στην αρχή της εντολής σας και ειδικότερα το 2011. Υπήρξε μια περίεργη αύξηση των επιτοκίων τότε και τώρα εκ των υστέρων πολλοί νομίζω θεωρούν ότι ίσως αυτό τότε να ήταν λάθος. Αν δείτε όμως και το επίπεδο του πληθωρισμού τότε, θα δείτε και από πού προήλθε αυτή η αύξηση των επιτοκίων. Σας ερωτώ λοιπόν, ρίχνοντα μια ματιά προς τα πίσω τελευταία 8 χρόνια και ειδικότερα αυτό το επεισόδιο, αν σκεφτείτε σήμερα τα επιτόκια, θα λέγατε ότι πρέπει να είμαστε μάλλον προσεκτικοί, διότι μιας και είμαστε σχεδόν στο μηδέν, μήπως θα έπρεπε να είμαστε προσεκτικοί ή θα λέγατε ότι τα διδάγματα του 2011 είναι να μην ανησυχούμε και τόσο πολύ για τα σημερινά επιτόκια που είναι σχετικά χαμηλά, αλλά για τι θα γίνει ίσως ε, δύο ή τρία χρόνια αργότερα. Πρώτη ερώτησή μου λοιπόν αυτή. Ίσως αυτό σας δώσει μια ευκαιρία να εξηγήσετε λίγο και πώς βλέπετε τα πεπραγμένα σας. Δεύτερη ερώτηση, μια παρατήρηση που κάνατε αρχικά σχετικά με το έντις. Αναφερθήκατε σε τρία ζητήματα για την μείωση του κινδύνου που ίσως θα πρέπει να έχει κανείς υπόψη του όταν πάει να συνάψει μια συμφωνία. Ένα που μου φάνηκε να λείπει ωστόσο είναι αυτό που έχει να κάνει με, το, με τον κίνδυνο του δημοσίου χρέους. Και διαρωτώ με εάν αυτό ε, το αφήσατε απ' έξω ε, λόγω χρόνου, δηλαδή αναφερθήκατε μόνο σε τρία σημεία και όχι σε τέσσερα, ή δεν θεωρείτε ότι αυτό το sovereign risk δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί στους ισολογισμούς των τραπεζών στα πλαίσια του έντις. Και η τρίτη μου ερώτηση αναφέρεται σε κάτι που διάβασα με ενδιαφέρον. Άλλωστε, ε, το Bloomberg φαίνεται πως στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μαρτίου, ε, της 21ης Μαρτίου αναφερθήκατε στο ε, πλαίσιο ρευστότητας για εξυγίανση τραπεζών και είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδεχομένω να προσφέρει ρευστότητα σε καλέ τράπεζε, εάν μπορέσει μία να προκύψει, αλλά ε, με χαμηλότερα στάνταρτ για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία. Αυτά λέει το δημοσίευμα του Bloomberg. Εσείς όμως ήσασταν παρόν στην συνεδρίαση για να σας διευκολύνω. Θα ρωτούσα, θεωρείτε ότι χαμηλότερα στάνταρτ για τα κολάτερα για τις εγγύσεις δηλαδή είναι καλές ή όχι. Είναι καλά ή όχι. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Για το επεισόδιο του 2011 και την αύξηση των επιτοκίων. Όπως είπατε, εκ των υστέρων Ρώμενο μπορεί να έχει κανείς διαφορετική άποψη για το επεισόδιο, αλλά πρέπει να τονιστεί ακόμη ότι την εποχή εκείνη μιλούμε για αλλαγές επιτοκίων λίγο πριν από το καλοκαίρι του 2011. Την εποχή εκείνη ο πληθωρισμός ήταν γύρω στο 2,5%. 2,7% στην Ευρωζώνη και η ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο ήταν γύρω στα 2%. Άρα οι εξελίξεις του πρώτου μισού του 2011 φαίνονταν να δείχνουν ότι η ανάκαμψη μετά από την κρίση του 2008-2009 είχε αρχίσει. Σας βάζω το πλαίσιο μέσα στο οποίο λήφθηκαν τότε οι αποφάσεις εκείνες. Βέβαια τα όσα συνέβησαν μετά, μετά το καλοκαίρι του 2011 δηλαδή, απέβησαν πολύ διαφορετικά από αυτά που είχαν γίνει στο πρώτο εξάμεινο του 2011. Όλες οι προβλέψεις οικονομικής ανάπτυξης αποδείχθηκαν εσφαλμένες, διότι η οικονομία επιβράδυνε σημαντικά και απότομα στο δεύτερο μισό του 2011 με τις επιπτώσεις στον πληθωρισμό και η κατάσταση εμφανίστηκε πολύ διαφορετικά. Και ως αποτέλεσμα αυτού πήραμε πίσω τις αυξήσεις αυτές το Νοέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Και όπως γνωρίζετε η νομισματική πολιτική πάντοτε έχει μια υστέρηση χρόνου και σημαντική μάλιστα μέχρι να αποδώσει. Κάνοντας αυτές τις αυξήσεις επιτοκίων εκείνους τους μήνες, δεν θα αποτελούσε εξήγηση για την δεύτερη ύφεση που αντιμετωπίσαμε το 2012 και 2013. Η εξήγηση για αυτή τη δεύτερη ύφεση βρίσκεται απολύτως μέσα στην δημοσιονομική πολιτική και η ταυτόχρονη δημοσιονομική εξυγίανση που αναλύθηκε από όλες τις χώρες μέρη της Ευρωζώνης στη διάρκεια εκείνων των ετών. Αυτά είναι άλλωστε τεκμηριωμένα και σε έγγραφα της Κομισιόν. Με μοντέλα που δείχνουν τα αποτελέσματα εκείνων των ταυτόχρονων δημοσιονομικών εξηγιάσεων. Τώρα ξαναλέω ότι εκ των υστέρων ορόμενα αυτά μπορούμε να πούμε ότι δεν επιβεβαιωθήκαν οι προβλέψεις που είχαν γίνει τότε, όμως κάναμε πολύ γρήγορα διορθώσεις στις ε, αυξήσεις εκείνες. Διορθώσαμε τις αυξήσεις εκείνες το ε, Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Τώρα για το sovereign risk, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όπως και η έκθεση των πέντε προέδρων. Η έκθεση των πέντε προέδρων αναγνωρίζει ότι υπάρχει εδώ ενδεχομένως ένα θέμα, διότι αν υπάρξει υπερβολική συγκέντρωση στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών εσωτερικού χρέους μπορεί σε περιπτώσεις στρες να οδηγήσει σε τροτότητα των τραπεζών. Όμως η έκθεση των πέντε προέδρων λέει ταυτόχρονα ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται και στα πλαίσια παγκόσμιας, διεθνούς αλλαγής της αντιμετώπισης του sovereign debt. Και αυτό θα πρέπει να το αποφασίσει η Επιτροπή της Βασιλείας ιδεμή θα έχουμε πρόβλημα ισο, ισο, ισότιμων όρων ανταγωνισμού. Το ερώτημα αυτό του κινδύνου δηλαδή του δημοσίου χρέους στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών είναι πολύ περίπλοκο και λόγω χρόνου δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Πολλά πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη και ιδίως το ότι η αδίποτε αλλαγή δεν θα πρέπει να οδηγεί αμέσως σε σημαντική αστάθεια σε κάποιες αγορές δημοσίου χρέους που αποτελεί ανησυχία, διότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχουν χώρες όπου κάθε χρόνο διαθέτουν δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πρέπει να αποπληρώσουν δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο ε, δημοσίου χρέους. Και για να μπορέσει να γίνει αυτό χωρίς μεγάλες αναταράξεις, βασίζονται βέβαια στους προηγούμενους κατόχους αυτών των ομολόγων τα οποία λήγουν. Αυτό είναι ένα πρόβλημα μεταξύ άλλων. Θα σας προτείνω να διαβάσετε το κείμενο της ομιλίας μου του Μαΐου που θα είναι το αποχαιρετιστήριο σε μια διάσκεψη της Κεντρικής Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που θα ε, διεξαχθεί τότε και εκεί θα αναφερθώ με περισσότερες λεπτομέρειες στο θέμα αυτό του ε, κινδύνου δημοσίου χρέους. Σε ό,τι αφορά την ρευστότητα στην εξυγένση, αυτή η είδηση που αναφέρατε ε, βρίσκεται σε κάποια σύγχυση, ακόμα και για το ίδιο το θέμα, διότι το θέμα δεν είναι βέβαια, δεν σχετίζεται με την προσφορά εξυγίανση στην καλή τράπεζα που θα προκύψει μέσα από την εξυγίανση. Εάν προκύψει είναι καλή τράπεζα. Good Bank έχει την ε, τραπεζική της άδεια λειτουργίας, ε, την εποπτεία της, είναι εξυγιασμένη και αν συμβαίνει αυτό έχει πρόσβαση σε δράσεις ε, νομισματικής πολιτικής όπως η οποιαδήποτε άλλη τράπεζα. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή δηλαδή σε ό,τι αφορά την καλή τράπεζα που προκύπτει μέσα από τη διαδικασία εξυγίανσης. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα πρόβλημα και καμία αλλαγή. Το δεύτερο θέμα είναι βέβαια ότι στη διαδικασία της εξυγένσης που μπορεί να χρειαστεί κάποιες μέρες, πολλές, λίγες, κάποιες μέρες. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, σε, αυτή την, ε, σε αυτό το χρονικό πλαίσιο και αν δεν υπάρχει moratorium, άλλο ευαίσθητο θέμα αυτό, αν όμως δεν υπάρχει moratorium στη διάρκεια της διαδικασίας εξυγένσης μπορεί να προκύψουν ανάγκες ρευστότητας της τράπεζας αυτής την ώρα ακόμα που εξηγένεται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι εξηγένση, δηλαδή, μάλλον δεν είναι ε, ρευστότητα για την καλή τράπεζα. Είναι για αυτή την σύντομη περίοδο. Και εδώ αναφέρομαι μονάχα σε αυτά που υπάρχουν ήδη και που έχουν ήδη αποφασιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και υπάρχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ηνωμένο, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο η Bank of England έφτιαξε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ένα μηχανισμό για να δίνει ρευστότητα στην εξυγίανση για εκείνες τις περιόδους χρόνου, για τις λειτουργίες εκείνες συγκεκριμένα. Γι' αυτό όμως η Τράπεζα της Αγγλίας θα λαμβάνει εγγύηση από τη Τσαυροφυλάκιο. Διότι βέβαια υπό ε, φυσιολογικές συνθήκες, και εμείς το σεβόμαστε απολύτως αυτό, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να προσφέρει ρευστότητα σε μια ευάλωτη τράπεζα ή η τράπεζα που βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης, γιατί αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα έχει δηλωθεί ως ε, κινδυνεύουσα να πτωχεύσει. Πρόκειται λοιπόν για ιδιαίτερη περίπτωση. Όμως Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν προβλέψει διαδικασίες που λέγουν ότι υπάρχει μια διαδικασία εξυγένσης που εφόσον προκύψουν προβλήματα αριστότητας, τότε ανταποκρίνονται και ελπίζω η Ευρώπη να φτάσει και η ίδια σε κάποια λύση στο πρόβλημα αυτό, που χρειάζεται πραγματικά τέτοια πρόβλεψη για να υπάρχει ένα πλήρες και στέρεο σύστημα εξυγέννησης των τραπεζών. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπερές. Ευχαριστώ εξ τους των σοσιαλιστών. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για όλες σας αυτές τις κριτικές παρατηρήσεις, διότι είναι τελευταία σας παρουσία εδώ ε, στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ και εγώ, παρόλο που το έκαναν και οι συνάδελφοι πριν από μένα. Να θέσω και εγώ δύο ερωτήσεις με τη σειρά μου. Η πρώτη έχει να κάνει με την έκθεση στην οποία είμαι συνεισηγήτρια με τον γείτονά μου ως, ε, και είναι και βοηθητικός θα έλεγα ως ε, εκπρόσωπος του ΕΛΚ για τις αρχές εποπτείας και τη δυνατότητα να καταρτήσουμε τεστ αντοχής, stress test θα μα πείτε εσεί, βέβαια αν γίνεται στο επίπεδο τη Τραπεζικής Ένωση, αλλά μα ενδιαφέρει και κατά πόσο είναι οι κλιματικοί κίνδυνοι, ε, οι κλιματικέ απειλές και τα διάφορα σενάρια που μπορούμε να καταρτήσουμε, θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη, γιατί για την ώρα δεν αποτελούν μέρο των ανησυχιών των ε, υπευθύνων των κεντρικών τραπεζών. Θα έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη στο επίπεδο των ε, stress test. Και η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τον τρόπο που η Κεντρική Τράπεζα τοποθετείται όταν εκφράζεται για τον διορισμό ενός από τα τελευταία μέλη, του, μέλη της. ο διορισμός του διαδόχου σας, όπως ξέρετε, ε, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων επικριτικών σχολείων, τα οποία ήταν και θεμητά. Διότι ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβόλου ε, είναι, ε, Συμβουλίου είναι μέρος της ε, νομιμοποίησης που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ λοιπόν είχαμε μια πολύ σύντομη γνωμοδότηση, χωρίς καμία επιχειρηματολογία, κανέναν δημόσιο διάλογο. Πιστεύετε ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να προχωρά ε, η Κεντρική Τράπεζα στο διορισμό. Με αυτή την πρακτική μπορεί να διαρκέσει ή θα μπορούσε κάτι να αλλάξει. Και η τελευταία μου ερώτηση που παραπέμπει και στην πρώτη, σε ό,τι αφορά την ε, ποσοτική χαλάρωση και την στρατηγική αυτή της αγοράς. Ε, για λόγους διαφάνειας από την πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας και για τους τίτλους που αγοράζονται. Είναι αρκετά τα όσα δημοσιοποιούνται, θα μπορούσαμε να πάμε και παραπέρα. Και με ποια στρατηγική δημοσιοποίησης. Διότι σε αυτές τις αγορές γίνονται αγορές και στο επίπεδο της brown οικονομίας, της πράσινης οικονομίας. Και όλα αυτά κάπως μπορεί να ε, εμπλέκονται στη στρατηγική που μπορεί άλλοι να προσπαθούν να κατακτήσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Και εδώ θα περάσω στα αγγλικά. Σε ό,τι τα τεστ αντοχής και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Όπως είπατε, οι περιβαλλοντικοί κινδύνοι, οι κλιματικές απειλές δεν συμπεριλαμβάνονται στα κλασικά τεστ αντοχής που γίνονται τώρα. Θα ήταν δύσκολο και συμφωνώ ότι θα χρειαζόταν και θα πρέπει να γίνει, είναι να έχουμε κάποια ευαισθησία στις αναλύσεις που κάνουμε για την καταμέτρηση των περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Εκεί είναι η μεγαλύτερη κίνδυνη και απειλές. Όμω τα σημαντικά περιβαλλοντικά ατυχήματα δεν μπορούν να αποτελέσουν μέρο ενό κλασικού, ενό επαναλαμβανόμενου τεστ αντοχή. Είναι κάτι το έκτακτο λόγω του βαθμού ε, των πιθανότητων. Ε, η Τράπεζα της Αγγλίας, λόγου χάρη, έχει προσπαθήσει να καταρτήσει ένα σενάριο για το τι θα γίνει αν ας πούμε κλιματικές αλλαγές και η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξήσουν τη στάθμη ε, των θαλασσών και πώς αυτό θα επηρέαζε τα περιουσιακά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτή είναι μια ευαισθησία συγκεκριμένη την οποία δεν μπορώ να πω ότι θα είναι εύκολο να τι περιλάβει κανεί ένα κλασικό τεστ αντοχή, αλλά καλό είναι να λυθεί υπόψη, γιατί σίγουρα υπάρχει απειλή για αυτά τα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία. Οι ίδιε οι τράπεζε, α πούμε, θα πρέπει να ανησυχούν για λόγου ασφαλιστικού και όλε οι ασφαλιστικέ εταιρείε. Ε, θα πρέπει να σκεφτούν αυτά τα πιθανά γεγονότα. Είμαι σίγουρο ότι οι ασφαλιστικέ εταιρείε τα σκέφτονται. Τα γνωρίζουν αυτά, αλλά καλό θα ήταν να περιληφθούν και στις μέρημνες των εποπτών για να δουν τι θα έκαναν σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη σας ερώτηση, δεν βλέπω τις διαδικασίες όπως προβλέπονται βάσει της νομοθεσίας να αλλάζουν, αλλά όπως ξέρετε αυτό είναι επιλογή του Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο και η ΕΚΤ απλώς ε, γνώμη δίνουν Αποφασίζει όμως το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οπότε εκεί δεν μπορώ να ε, προβλέψω κάποια αλλαγή. Και σε ό,τι αφορά την τελευταία σας ερώτηση, ναι, έχει εκφραστεί περιέργεια και έχουν τεθεί ερωτήσεις για τα προγράμματα αγοράς υπό αυτήν την σκοπιά και κατά πρώτον να πω ότι υπήρξαμε πλήρως διαφανείς ό,τι αφορά τα προγράμματα αγορών μας. Σε ό,τι αφορά και τα κρατικά ομόλογα, όπου δώσαμε πλήρη ενημέρωση και μάλιστα έχουμε δώσει και προβλέψει για το ποιε πιστεύουμε ότι θα είναι οι αποπληρωμέ και οι εξηγιάνσει, οι εξαγορέ μέχρι το τέλο τη χρονιά. Τώρα για τα εταιρικά ομόλογα. Είμαστε κεντρική τράπεζα που δίνει τις περισσότερες πληροφορίες σε σύγκριση με την οποιαδήποτε άλλη κεντρική τράπεζα έχει αγοράσει κρατικά ομόλογα. Και εταιρικά μάλλον ομόλογα όχι απλώς δίνουμε τα ποσά, δίνουμε και τον κατάλογο των συνολικών ποσών, δηλαδή δίνουμε λεπτομερή στοιχεία για το πώς καταλήγουμε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο. Καμιά άλλη κεντρική τράπεζα δεν το έχει κάνει αυτό. Και απλώς δεν αποκαλύπτουμε πόσο κάθε κεντρική τράπεζα έχει αγοράσει από κάθε αξιόγραφο. Γιατί, γιατί μας απασχολεί να γίνονται οι αγορές έχοντας κατά νου το νομισματικό αντίκτυπο που θέλουμε να πετύχουμε, κάνοντας ακριβώς αυτές τις αγορές, αλλά δεν θέλουμε να πλεχτούμε στην διαμόρφωση των τιμών στην αγορά. Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι οι επενδυτέ, οι εταιρείε και οι τράπεζες θα ήθελαν να ξέρουν ακριβώς ποιο αγοράζει τι και πόσο από το κάθε ομόλογο έχει κάθε κεντρική τράπεζα, γιατί άμα το ξέρανε, ε, και υπολογίζαν και την ορίμανση, θα μπορούσαν να κάνουν τους υπολογισμούς τους για το κέρδος ανάλογα με την κάθε περίοδο. Προφανώς τους ε, συμφέρει να ξέρουν τα πάντα. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε τέτοιες πληροφορίες που απλώς θα ε, κατέληγαν να επηρεάσουν τη δημόρφωση των τιμών, χωρίς να δίνουν κανένα άλλο ε, όφελος. Δίνουμε πολλά, πιστεύω ήδη. Για τα ομόλογα που αγοράζουμε, ε, ενημερώνουμε ποια αγοράστηκαν και ποια είναι τα συνολικά ποσά. Τώρα, από τα ομόλογα αυτά, έχουμε 47 πράσινα. 47 εκδόσεις πρασίνων ομολόγων. 5% του συνολικού χαρτοφυλακίου αυτού που έχουμε αγοράσει συνολικά. Παρόλο που αυτά τα 47 πράσινα είναι μόνο 3,8% του συνολικού ε, ποσού ομολόγων που αγοράζουμε. Όπως ξέρετε επίσης, Στηρίζουμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία έχει πολύ σημαντική δράση στην έκδοση των πρασινών ομολόγων. Αυτό για να τονίσω ότι δεν πρόκειται για ένα θέμα που το έχουμε παραβλέψει και θεωρώ ότι αυτό που κάναμε ήταν και το ε, ορθόν, χωρίς να θέτουμε να τους νομισματικούς σκοπούς του προγραμματό μας. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μπορούσατε να κάνετε το ίδιο και μεταξύ των εταιριών ε, ε, στοιχημάτων. Πάντως θα συνεχίσουμε την όλη συζήτηση και με τον υποψήφιο για τη θέση του Αντιπροέδρου για να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει βελτίωση στη διαφάνεια και σωστή τοχοθεσία. Στοχοθεσία στην αγορά των ομολόγων και των αξιογράφων είναι κάτι που θα μας απασχολήσει. Έχουν υποθεί πολλά για το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ήταν μια πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων αυτή που είχαμε. Ευχαριστούμε για την ποιότητα και το σοβαρόν της ε, προσπάθειας σας να απαντήσετε. Μπήκατε στην ουσία των πραγμάτων και πάντοτε εκτιμούμε αυτήν σα την στάση ε, όταν έρχεστε και συζητάμε. Ευχαριστώ και πάλι, Αντιπρόεδρε Κωνσταντζη, ευχαριστούμε για, την, ε, ε, για τις που προσφέρατε στο Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την θέση σας. Νομίζω ότι αξίζεται και ένα χειροκρότημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι η μετεκατάσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Καθορισμός της έδρας, έχουμε τις τροπολογίες, που είναι οι εισηγητές μας. Είναι απλό το θέμα, δεν χρειάζεται να κάνουμε εισαγωγή. Έχουμε τις τροπολογίες να εξετάσουμε στην έκθεση αυτή, Μπάλτς και Μπέρες. Οπότε θα δώσω το λόγο στους συνεισηγητές. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριος Μπάλτς. Ευχαριστώ που προβλέψατε την ανταλλαγή απόψεων για τις τροπολογίες είναι περιορισμένο ο αριθμός των τροπολογιών. Συνολικά είναι 19. Από τη δική μου σκοπιά θα ήθελα να υπενθυμίσω πρώτα τα βασικά της κοινή αυτή προτάσεω ψηφίσματο της Περβάνος Σουμπερέ και δική μου για την μετεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής τα βασικά είναι τα εξή. Αφενό η κριτική που έχουμε ασκήσει στον τρόπο που λήφθηκε απόφαση από Συμβούλιο και Επιτροπή. Δεύτερο, η αξίωσή μα να λάβουμε περισσότερε πληροφορίε για το πώ ελήφθη η απόφαση αυτή και ιδίω ποια ήταν τα κριτήρια για τη λήψη αποφάσεως. Τρίτο, η άλλη αξίωσή μας για την επανεξέταση της κοινή δήλωσης για τους ε, οργανισμούς όπως πάντοτε δήλωσε το Κοινοβούλιο. Τέταρτο, σαφής υπενθύμηση ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει εξουσίες συνομοθέτου στο ζήτημα της, ε, του ορισμού της έδρας. Εξάλλου, θέλουμε να διατηρήσουμε τις αρμοδιότητες ε, της, τρα, της τραπεζικής ε, εποπτικής αρχής, ανεξαρτήτως της μελλοντική έδρας. Και τέλος, θα θέλαμε να έχει προετοιμαστεί και να είναι έτοιμη η μετεγκατάσταση, η μετακίνηση της τραπεζικής εποπτικής αρχής μέχρι την αποχώρηση του, μεγάλου, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτά τα βασικά δεν αμφισβητούνται από τις τροπολογίες που έχουν κάνει οι συνάδελφοί μας. Όπως είπα υπάρχουν μόνο 19, 19 τροπολογίες επί του νομοθετικού ψηφίσματος είναι η αριθμή 5 έως 19, διορθώνει η κυρία Μπερές δίπλα μου και το ξεκαθαρίζω. 5 έως 19, άρα συνολικά είναι 14 Έχουμε λοιπόν μόνο 14 τροπολογίες για το νομοθετικό ψήφισμα και πάλι από αυτές τις 14 δεν αναφέρονται όλες στην μετεγκατάσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εποπτείας Τραπεζών. αναφέρονται σε ποιότητα και ποσότητα της ε, ρύθμισης ε, των ε, χρηματοπιστωτικών μετά από το Brexit. Η δική μου πολιτική ομάδα, το Λαϊκό Κόμμα, δεν έχει υποβάλει καμία τροπολογία. Δηλώνω εδώ και πάλι την υποστήριξη της πολιτικής μου ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο, στην πρόταση ψηφίσματος. Δηλαδή θα θέλαμε να υπάρξει δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αναθεώρηση της κοινή δήλωση των δύο άλλων θεσμικών οργάνων, όπως κάναμε και για τον οργανισμό φαρμάκων. Στην περίπτωση αυτή θα θέλαμε να εγκαταλειφθούν οι εθνικοί εγωισμοί και να παίξουμε το θεσμικό μας ρόλο. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξεκαθαρίσουμε ότι απόφαση χωρίς συμμετοχή του Κοινοβουλίου δεν είναι δυνατόν να ληφθεί. Στις 24 Απριλίου θα πρέπει να ψηφιστεί το κείμενο για να μπορέσει το δυνατόν συντομότερο να αρχίσει ο τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπερές. Ε, ευχαριστώ πολύ. Τα είπε και ο Μπούχαρτ τα κύρια σημεία. Δεν θα επανέλθω στην πρόταση των συνεισηγητών. Έχει ήδη συζητηθεί. Τώρα για τις 14 τροπολογίες που υποβλήθηκαν. κάποιες τις υπέβαλαν σοσιαλιστές. Εννοείται ότι συμφωνώ με τις περισσότερες από αυτές. Ίσως όχι με όλες. Όλος παραδόξους. Πάντα το βασικό εδώ είναι να διατηρήσουμε το πνεύμα της πρότασης των συνεισηγητών. Και ποιο είναι αυτό το πνεύμα. Είναι αυτή η μετεγκατάσταση, αυτή η μεταφορά της Ευρωπαϊκής, Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ε, να γίνει κατά από καλές συνθήκες και όπως το ζητά και η Επιτροπή Προϋπολογισμών στο κάτω-κάτω με κέρδος τελικά δημοσιονομικό ή δυνατόν. Και κυρίως να αποφεληθούμε από αυτή την ευκαιρία για να υπενθυμίσουμε ποιος είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε τέτοιου είδου περιστάσεις. Υπάρχει κοινή δήλωση του 2012, αλλά προφανώς δεν είναι προσαρμοσμένη στην σημερινή κατάσταση. Αλλά θέλω ε, να προσθέσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει το άνοιγμα της δήλωσης αυτής πάλι, γιατί θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από τη λήξη της θητείας να δημιουργηθεί μια νέα, ένας νέος οργανισμός, δεν ξέρω με τι όνομα, Πάντως υπάρχει πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία ενός οργανισμού για την εργασία, ας πούμε, ε, που θα εποπτεύει τις εθνικές ε, επιθεωρήσεις εργασίας. Πώς θα παρεύει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα κριτήρια προκειμένου να αποφασιστεί η έδρα αυτής της νέας αρχής. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Για μένα το σημαντικό είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα να αρχίσει η συζήτηση με το Σεβούλιο για να σταθεροποιηθεί το νομικό πλαίσιο αυτής της μεταφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών γιατί πέρα από το πολιτικό σκέλος χρειάζεται και μια ολόκληρη πρακτική δομή. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι χρειαζόμαστε από την πρώτη μέρα να μπορεί να αρχίσει στη νέα της έδρα η υπηρεσία αυτή. Ε, να μην εξετάσω τώρα μία-μία τις τροπολογίες, πάντως μπορούμε να τις υποστηρίξουμε Υπάρχει μία που νομίζω ότι είναι απαράδεκτη, Πρόεδρε, γιατί αμφισβητεί την ίδια την συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα άλλα, να συμφωνήσω βέβαια με τον συνεισηγητή μου για να δω που θα κατευθυνθούμε τελικά. Αυτό όσον αφορά τις 14 τροπολογίες που υπέβαλαν οι συνάδελφοι και υπάρχουν και άλλες 5 βέβαια που έχουν υποβάλει οι συνεισηγητές. Τώρα για τις νομοδοτήσει των δύο άλλων επιτροπών προϋπολογισμών και συνταγματικών υποθέσεων. Ε, για τη δεύτερη περίπτωση είναι κάπως πρωτότυπη η αντίδραση της Επιτροπής αυτής, γιατί την πρωτοβουλία του συναδέρφου μας Έλμαρ ε, Μπροκ ενέκρινε δήλωση η οποία προσαρτίστηκε στην ψηφοφορία που έγινε για τη νέα έδρα της, του Οργανισμού για τα Φάρμακα. Και είναι καλό για τη συνέπεια να ακολουθήσουμε το ίδιο, αλλά μπορεί να είναι περιττό δεδομένο των όσων έχουμε ήδη εμείς. Δεν χρειάζεται να πούμε δηλαδή τρεις φορές τα ίδια πράγματα, ότι το κοινοβούλιο πρέπει να εισακούεται. Για να το πετύχουμε πρέπει να είμαστε συνεπείς. Τώρα, για την Επιτροπή Προπολογισμών, οι τροπολογίε τους είναι προτάσει όχι μόνο στην ομοθετική πρόταση, αλλά και στην πρόταση ψηφίσματος. Και νομίζω ότι περισσότερες από αυτέ θα έπρεπε να υιοθετηθούν από την Επιτροπή μας. Πάνε προ τη σωστή κατεύθυνση προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σανταλούντς. Εσείς κύριε Λούκα. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ τον κύριο Λούνες που ε, κολλείεται σήμερα. Με παρακάλεσε να διαβάσω την εξής δήλωση εξ ονόματός του. Συμφωνούμε με τη γενική διατύπωση του σχεδίου του Λαϊκού Κόμματος Υποστηρίζουμε δύο τις παρατηρήσεις που γίνονται όσον αφορά την σχέση μεταξύ EBA και ESMA, το ίδιο και για την διαδικασία ψηφοφορίας. Υπάρχει ένα ακόμη σχόλιο, ωστόσο, που επιθυμώ να κάνω, λέει ο συναδελφό μου, και το έχω κάνει στι τροπολογίε μου, διότι οποιαδήποτε αναθεωρημένη δήλωση για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και οποιοδήποτε ενισχυμένο ε, ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα προβλέπονται στα, ε, στη δήλωση αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την γεωγραφική ισορροπία και την ισορροπία μεταξύ μεγάλων και μικρών χωρών. Η γεωγραφική κατανομή και οι ενδεχόμενες ενδεχόμενα μειονεκτήματα για τις μικρότερες χώρες έχει ήδη το, ε, γίνει από τον κύριο Χέις σε παλαιότερη τοποθέτηση. Υπάρχουν ε, χώρες μέλη που ακόμη δεν διαθέτουν έδρα οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ήμασταν ευγνώμονες αν οι συνεισηγητές μπορούσαν να το λάβουν υπόψη τους αυτό στην τελική τους έκθεση. Αυτά λέει ο κύριος Λούνης, ο οποίος εν τέλει ευχαριστεί. Ευχαριστώ εσείς κύριε Κλίντς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με την έκθεση και με τα σχόλια ε, του συναδέλφου μου Μπάλτς Πράγματι θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβουμε και να παίξουμε τον θεσμικό μας ρόλο χωρίς ναι μεν αλλά. Και οφείλω να σημειώσω ότι τα τελευταία χρόνια το Συμβούλιο δεν έχει αφήσει να του φύγει ευκαιρία για να τονίσει με τη στάση του ότι θεωρεί ότι είναι τουλάχιστον ανώτερος μεταξύ ίσων, πρώτος μεταξύ ίσων, να το πω καλύτερα για να μην πω και τίποτε χειρότερο. Χρειάζεται λοιπόν να μιλήσουμε και εμείς με καθαρή γλώσσα. Το γεγονός ότι τόσο η EBA όσο και η ε, SMA λαμβάνουν την τελική του έδρα όπως τη λαμβάνουν, δείχνει, μου δείχνει ότι τα κριτήρια επιλογής δεν είναι σαφή. Εάν είναι σαφή τα κριτήρια επιλογής και διαφανή και τα οποία δύναται κανείς να συζητήσει καθαρά και δημόσια, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να μπορεί να καταλήξει και σε μια ε, λίγο πολύ ομόφωνη απόφαση και να μην χρειάζεται προσφυγή σε κλήρωση. Μου φαίνεται λοιπόν πολύ ατυχή η λύση αυτή και παρόλο που είμαι Γερμανός Ευρωβουλευτής θα προτιμούσα ε, να είχε σταλεί η EBA σε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης, για παράδειγμα Σλοβακία. Η Πρατισλάβα άλλωστε είχε ζητήσει να λάβει τη θέση του οργανισμού, την έδρα συγγνώμη, του οργανισμού αυτού. Εγώ θα προτιμούσα πράγματι να ε, λάβει την ε, ε, έδρα αυτή η Μπρατισλάβα. Μπορώ να συμφωνήσω με τον Λούνες που μίλησε προηγουμένως διαστόματος του συναδέλφου μας που ήδη αποχώρησε βέβαια για τη γεωγραφική κατανομή αλλά δεν μπορώ να συμφωνήσω εκεί που λέει ότι όσο μεγαλώνει ο ρόλος του Κοινοβουλίου, τόσο μειώνεται η βαρύτητα των μικρών χωρών μελών. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με τη δήλωση αυτή και γι' αυτό δεν θα υποστηρίξω την τροπολογία του υπαριθμού 13. Επίσης ε, με ενοχλεί η τροπολογία 14, τάνκ, διότι δυνατόν είναι οι backup services μεταξύ SMA και EBA να γίνει pool, να γίνουν σε pool, δηλαδή σε δεξαμενή κοινή, όχι όμως μεταξύ τριών ε, οργανισμών. Εγώ λοιπόν εκεί προτιμώ το κείμενο του αρχικού ψηφίσματος, του αρχικού σχεδίου ψηφίσματος. Εν τέλει, συμφωνώ με την έκθεση, με εξαίρεση δε των δύο αυτών τροπολογίων που μόλις ανέφερα, συμφωνώ και με τις κατατηθείς τροπολογίες. Ευχαριστούμε. Σε κάθε περίπτωση η Σλοβακία είχε ζητήσει τον οργανισμό φαρμάκων, οπότε δεν μπορεί να θέσει πάλι υποψηφιότητα. Ευχαριστούμε όμως Φέν Κίλκολτ. Ναι, δεν υποβάλαμε τροπολογίες, διότι πολύ απλά μας ικανοποιεί το σχέδιο έκθεσης. Οπότε, έχοντας διαβάσει όλες τις τροπολογίες, δεν είμαι καθόλου πεπισμένος ότι καμία από αυτές είναι απαραίτητη θα μπορούσαμε απλώ να ψηφίσουμε την έκθεση ω έχει, αλλά μπορούμε να δεχτούμε και κάποιε τροπολογίε. Δεν κάνονται καμιά συγκλονιστική διαφορά. Κάποιε με παραξένεψαν, αλλά τέλο πάντων δεν είναι επί τη ουσία. Η ουσία του θέματο για μένα είναι ότι θεσμικώ λέμε ότι είναι λίγο περίεργο να έχουμε δύο αποφάσεις με κλήρωση και ότι το Συμβούλιο δεν έχει λάβει πολύ σοβαρά υπόψη το γράμμα του νόμου. Ένα παρόμοιο πρόβλημα είχαμε και στο επίπεδο των διορισμών στην ΕΚΤ, όπου είδαμε να υπάρχουν κάποιε θεσμικέ διαφωνίε. Αντί λοιπόν να τα λέμε μεταξύ μα, καλό θα ήταν να ενημερώσουμε το κοινό για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και με το Eurogroup για τους διορισμούς στην ΕΚΤ. Διότι βλέπω εδώ να υπάρχει μια παράλληλη διαδικασία, ένα παράλληλο πρόβλημα. Ποιος είναι ο ρόλος του δικού μας σώματος όταν ε, φτάνουμε στο επίπεδο μιας συζήτησης όπου καταλήγουμε να έχουμε το Συμβούλιο να θεωρεί ότι μπορεί να αποφασίσει μόνο του. Και αν έχουμε διαφορετικές απόψεις επί ενός συγκεκριμένου θέματος, τελικά πόσο σοβαρά λαμβάνουν την απόψή μας. Αυτό έχει να κάνει και με το πόσο σοβαρά λαμβάνουμε εμεί οι ίδιοι τον εαυτό μα και τον ρόλο μα. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Πέραν αυτού, ελπίζω να έχουμε μια σύντομη ψηφοφορία επί τη συγκεκριμένη έκθεση. Ευχαριστώ. Θα σα απαντήσω εγώ, αλλά. Μαρίζα, εκ μέρου του κ. Παδημούλη. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Δεν μπορεί να είναι εδώ ο κ. Παπαδημούλη, οπότε εκ μέρου του ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο εισηγητέ για τη δουλειά τους και θα διαβάσω τη δήλωσή του. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό, το Κοινοβούλιο ήθελε να διευκρινίσει κάποια πράγματα, ιδίως ό,τι αφορά την δικασία λήψη αποφάσεων. Ως ομάδα επανειλημμένως έχουμε υπογραμμίσει ότι αυτές οι συμφωνίες σε σχέση με την έδρα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εποπτείας είναι κάτι για το οποίο θέλω να έχουμε άποψη. Αυτό που πρέπει να διασφαλίσουμε όμως σήμερα είναι ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για, την, ε, για τον καθορισμό της έδρας της ε, ΕΑΤ. Εδώ λοιπόν θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα γίνουν σεβαστές όλες οι ανάγκες και των εργαζομένων της. Θα πρέπει να υπάρχει μια έντιμη και ειλικρινή συνεργασία σε όλη τη διάρκεια του νομοθετικού κύκλου για να υπάρχει και ποιοτική τοποθέτηση των συνομοθετών. Και αυτά τα ορίζει και το άρθρο 295 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μα για το γεγονό ότι ο καθορισμό τη έδρα ε, συμφωνήθηκε μόνο με μια ε, ψηφοφορία μεταξύ των κρατών μελών. Θα πρέπει να υπάρξει ίση και ισότιμη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στην όλη διαδικασία και γι' αυτό θα θέλαμε να ξεκινήσει ε, άμεση αναθεώρηση τη κοινή δήλωση το 2012 για του αποκεντρωμένου οργανισμού Επίσης, δίνουμε μεγάλη σημασία στο κριτήριο της γεωγραφικότητας και της γεωγραφικής ισορροπίας σε σχέση με τον καθαρισμό των εδρών των οργανισμών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να υπάρξει καλή λειτουργία της ΕΑΤ θα πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένη η αρχή αυτή η δουλειά και οι συνθήκε εργασία των εργαζομένων, η ε, καλή του διαβίωση καθώ και αυτών των οικογενειών του είναι σοβαρά κριτήρια, το ίδιο με τα δημοσιονομικά και την διοικητική δυνατότητα και αποτελεσματικότητα. Η αμεροληψία και αξιοπιστία επίση τη ΕΡΤ είναι ε, ύψη τη σημασία. Γι' αυτό ε, θέλουμε τα ζητήματα αυτά να συζητηθούν περαιτέρω με τι συνεδριάσει των εισηγητών στο ερχόμενο διάστημα. Ευχαριστούμε ο κύριο Μονό. Δεν έχω σχόλια, πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καλώς. Ο πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στους συζητητές, αν θέλουν. Εγώ πρέπει να πω ότι συμφωνώ ότι έτσι κι αλλιώς αυτά που έπρεπε να πούμε λέγονται μέσα στην έκθεση, στο κυρίως σώμα της, του κειμένου. Συμφωνώ. Τώρα βέβαια και αυτά που λένε τροπολογίες καλές είναι. Η μόνη παρατήρηση που θα είχα να κάνω είναι αυτό που αναφέρεται εδώ ότι αποφασίστηκε στην παράγραφο 4. Οι χώρες μέλη δηλαδή αποφάσισαν μεταξύ τους η απόφαση όμως πρέπει να είναι αυτή, όχι αυτό που λένε εκείνες ότι αποφασίστηκε ήδη. Θα έλεγα δηλαδή ότι εδώ λείπει κάποια συνέπεια. Η Επιτροπή βέβαια κάνει μια πρόταση βάσει της απόφασης των χωρών μελών που δεν είναι σαφές εδώ αν πρόκειται για απόφαση του Συμβουλίου ή για απόφαση των χωρών μελών. Αλλά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανεξαρτήτως, τη κάνει την πρότασή της. Αλλά με συναπόφαση πρέπει να αποφασιστεί. Άρα εμείς μπορούμε να αποφασίσουμε αλλιώς, άμα θέλουμε. Εδώ συμφωνούμε μεν με το περιεχόμενο, αλλά δεν συμφωνούμε με τη διαδικασία. Αυτό είναι το ζήτημα. Τέλο πάντων, η έκθεση είναι καλή. Και για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή ρωτήσατε, το Κοινοβούλιο έστειλε επιστολή στον κύριο Τούσκ με αντέγραφο στον κύριο Σεντένο και την Προεδρία του Συμβουλίου και περιμένουμε απάντηση. Αν δεν έρθει η απάντηση, Θα το συζητήσουμε οι συντονιστές για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Είναι στο δικό μας χέρι τώρα. Λοιπόν, οι συγκητές. Η κυρία Μπερές. Και ο κύριος Βάλτς πιστεύει ότι όλα είναι εντάξει. Και εγώ στηρίζω πολλά από αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, ότι η αρχική πρόταση των συνεισηγητών ήταν η σωστή. Η μόνη μου επιφύλαξη είναι η πρόταση από την ΑΦΚΟ και τους προπολογισμού που πρέπει φυσικά να συμπεριλάβουμε στο τελικό σχέδιο. Και έτσι μπορούμε, πιστεύω, να έχουμε εντολή από την Επιτροπή να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πρόεδρος. Και εγώ καταλαβαίνω ότι η δηλώση ευθυγραμμίζεται με την έκθεση. Εσείς θα δείτε πώς θα συντονίσετε το όλο θέμα. Καλώς. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει 24 Απριλίου να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και στις 2 Μαΐου θα προχωρήσουμε με τις, ε, την απόφαση για τις διαπραγματεύσεις. Επόμενη συνεδρίαση, Δευτέρα 23 Απριλίου το απόγευμα και ολόκληρη την επόμενη μέρα την Τρίτη. Έλξη συνεδρίαση. Ευχαριστώ.